Αρχίζει τώρα η συνεδρίαση. Πριν προχωρήσουμε στην ακρόαση, υπάρχουν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως 11 και 12 που νομίζω ότι μπορούμε να διεξέλθουμε γρήγορα. Το 11 είναι το θέμα των κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοεφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών. Ξαναλέω λοιπόν, εισαγωγή ορισμένων κλωστών εμφαντουργικών προϊόντων. Την έκθεση Βαλέσα την έχουμε ήδη ακούσει. Πρόκειται για απλοποίηση του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως μπορεί να γίνει δεκτός έχει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να λάβει το λόγο. Όχι. Η Προεδρία του Συμβουλίου ίσως. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ε, ε, η Επιτροπή για τα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα σε 7 Φεβρουαρίου εξέτασε την πρόταση, δεν υπήρξαν σχόλια, εγκρίθηκε χωρίς ε, αλλαγές μετά από τη θετική ψηφοφορία ε, στην δική σας την Επιτροπή. Είναι έτοιμο το θέμα για κορεπέρ. Ωραία, οι σκιώδεις Πρόεδρε, νομίζω δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα που μένει να πούμε. Από διαδικαστικής πλευράς ε, υποστηρίζουμε το αίτημα του ΕΛΚΑ για την απλοποιημένη διαδικασία. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λούες. Δεν θέλετε, Μαρίκε. Ούτε Δεν έχω άλλον κανένα να ρωτήσω αν επιθυμεί να λάβει το λόγο. Ώστε κλείνει το θέμα αυτό. Προχωρώ στο θέμα υπαριθμών 12. Ψηφοφορία μόνο για την εκθέση αυτή. Όμως χρειαζόμαστε τις κάρτες ψηφοφορίας. Ελπίζω όλες και όλοι να τις έχετε. Ο Lightfried την έχει ξεχάσει. Πω πω πω πω. Είστε όλοι έτοιμοι. Αρχίζει η ψηφοφορία. Και ο κύριος Ρέν έχει ξεχάσει την κάρτα του και ο Σόλτς επίσης. Τρεις λοιπόν βουλευτές είναι υπέρ χωρίς κάρτες. Τέλος. Ναι, μάλλον έχει αρχίσει τώρα. Έκλεισε, τώρα τελείωσε. Άρα 22 ψήφισαν υπέρ, συν 3 χωρίς κάρτα, 25 λοιπόν και καμιά αποχή και καμία ψήφος κατά. Σας ευχαριστώ. Θέμα 13. θέμα για τις διαπραγματεύσεις για πολυμερή συμφωνία περί υπηρεσιών. Ο συνήθως είναι και ακρόαση αυτή δημοσία και μάλιστα μεταδίδεται και από το διαδίκτυο έτσι ώστε το κοινό που ενδιαφέρεται να μπορεί να παρακολουθεί. Θα διεξαχθεί στην βάση δύο πάνελ. Το πρώτο θα ασχοληθεί περισσότερο με μια οριζόντια ανάλυση των διαπραγματεύσεων και το δεύτερο θα εγκύψει σε ειδικότερους τομείς των υπηρεσιών Έχουμε και εκπροσώπους των συνενδιαφερομένων επιτροπών. Βλέπω τον κύριο Κοχ από την Επιτροπή Μεταφορών και ο κύριος Σάλμπα θα έπρεπε να είναι παρόν από την Οικονομική Επιτροπή, τον οποίον δεν βλέπω για την ώρα. Περνούμε τώρα στην ουσία της ακροάσεως. Ως γνωρίζετε, 24 χώρες στα πλαίσια των συνομιλίων της Γενέβης που επελέγει επίτηδες ως έδρα των συνομιλίων αυτών για να μην ε, είμαστε μακριά από τον ΠΟΕ συνδιαπραγματεύονται για μια περαιτέρω απελευθέρωση του τομέα των υπηρεσιών. Έχουμε ιδρύσει και μια ομάδα παρακολούθησης, monitoring group, που παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος πολύ προσεκτικά. Χαίρομαι που έχουμε και την διαρκή εισηγήτρια της Monitoring Group, κυρία Ρέντινγκ, είναι κοντά μας και της δίνω αμέσως τον λόγο για να κάνει μια σχετική εισαγωγή. Στα αγγλικά, κύριε Ρέντινγκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε ως εισηγήτρια για την ΤΙΣΑ. Έχω τρία προκαταρκτικά σχόλια να κάνω πρώτα, πριν να παραδώσω το μικρόφωνο στους πανελίστ. Πρώτο, η ΤΙΣΑ είναι ίσως η πιο σημαντική εμπορική συμφωνία που έχουμε διαπραγματευτεί ποτέ. Είναι ευρύτατη, άρχισε η διαπραγμάτευση τον Απρίλιο του 2013 και ε, σε συμφωνία με χώρες που θέλουν να προχωρήσουν σε περισσότερη απελευθέρωση του εμπορίου θα ε, συνδιαπραγματευόμεθα. Σε, με 24 χώρες μέλη του ΠΟΕ που είναι δηλαδή το 1 τρίτο των μελών του ΠΟΕ 70% δε ε, του συνολικού εμπορίου υπηρεσιών ανά τον κόσμο. Η ΤΙΣΑ είναι όπως είπα τη συμφωνία και συμπεριληπτική σε πολλούς, επεκτείνεται σε πολλούς τομείς όπως οι οικονομικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο, μεταφορές, η παρούσα νομική βάση ΚΑΤΣ έχει δημιουργηθεί από το 1995 και ε, επομένω πριν από την εποχή του διαδικτύου και πρέπει να ενημερωθεί. Είναι μοναδικέ αυτέ οι διαπραγματεύσει όσον αφορά και το εύρο του και την πολιτική του και η οικονομική του βαρύτητα. Άρα όλοι θα πρέπει να έχετε υπόψη σα την τίσα, να την βλέπετε στο ραντάρ σα δηλαδή. Και βεβαίω χρειάζεται και από την αρχή πλήρη διαφάνεια για να αποτραπούν οι εισδήποτε υπόνοιε, να διαλυθούν οι εισδήποτε μύθοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως εξήγησε ο πρόεδρος ήδη, έχει ιδρύσει μια ομάδα παρακολούθησης από τον Σεπτέμβριο ήδη του 2014 για να ενημερώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για να συνδιαμορφώνει τις διαπραγματεύσεις. Πρόκειται για έναν διάβλο ανοιχτό και από τις δύο πλευρές μεταξύ Κομισιόν και Κοινοβουλίου. Όμως οι συζητήσεις ε, διεξάγονται και πέραν από το Κοινοβούλιο και γι' αυτό έχουν ζητήσει από το Συμβούλιο να δημοσιοποιήσει την εντολή έτσι ώστε και ο υπόλοιπο κόσμος να μπορεί να γνωρίζει ακριβώς τι επιθυμεί η ευρωπαϊκή διαπραγματευτική πλευρά. Δεύτερο σχόλιο, η ΤΙΣΑ δεν πρέπει να πάρει τη μορφή της TTIP, ας το έτσι. Δηλαδή, από την αρχή χρειαζόμαστε μια επικοδομητική συζήτηση, έτσι ώστε να φύγουν από την τράπεζα διαπραγματεύσεων πράγματα που δεν θέλουμε και να μπουν μόνο πράγματα τα οποία πραγματικά επιθυμούμε. Όπως τα γνωρίζετε, ήδη από τον Ιανουάριο σε συνέντευξη τύπου κατέθεσα 10 κιανές και ελευθερές γραμμές έτσι ώστε να ε, απεμπλακούν τα δύο αυτά θέματα. Το ένα είναι για δυναμικό ανάπτυξης στην Αλοδαπή και το άλλο είναι για ενδεχόμενους ε, ευαίσθητους τομείς στην ημεδαπή. Το ένα είναι για τις ευκαιρίες και το άλλο είναι για τις ενδεχόμενες απειλές. Το ένα λοιπόν καλάθι περιλαμβάνει τα ερωτήματα, τα ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν διαμακρών και εις βάθος και το άλλο θα περιλαμβάνει τα πράγματα που δεν πρέπει καν να τεθούν υπό συζήτηση. Για να πετύχει η ΤΙΣΑ πρέπει να γνωρίζουμε σαφώς τι θέλουμε να πετύχουμε. Και μπορώ να σας δώσω και ορισμένα παραδείγματα. Μείωση των μη δασμολογικών φραγμών. Δημιουργία ενός πεδίου ισότιμου ανταγωνισμού σε ε, οικονομικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες να προσφερθούν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα στους καταναλωτές, για παράδειγμα, με την περιαγωγή, ε, να δοθεί πρόσβαση στις συζητήσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον βεβαίω δέχονται τους συμφωνημένους κανόνες, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η μελλοντική πολυμεροποίηση. Έχουμε και το ενδεχόμενο η Κίνα να μπει κάποια στιγμή στις διαπραγματεύσεις. Το άλλο που με απασχολεί είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα και για να πετύχει η ΤΙΣΑ πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς και τι δεν θέλουμε μεταξύ άλλων για τις δημόσιες υπηρεσίες, οι κοινοφελείς υπηρεσίες. Δεν θα πρέπει να μπουν στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Το, τα ρυθμιστικά δικαιώματα των κρατών, προστασία δεδομένων. Έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες που αποτελούν την βάση για τα πράγματα αυτά και δεν θέλουμε να θυγούν τα κοινωνικά στάνταρτ, να μην μειωθούν. Αυτά λοιπόν θα πρέπει άνευ καμιά αμφιβολία να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογή και να είμαστε απόλυτα σαφεί. Τα στοιχεία αυτά που ανέφερα είναι θεμελιώδη κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αδιαπραγμάτευτα. Έτσι, οι διαπραγματεύσεις ΤΙΖΑ θα πρέπει να υπακούν στις αρχές, για παράδειγμα του ΑΒ21 της συνθήκης μας, για την προστασία των θεμελιωδών αξιών, ελεύθερου εμπορίου, ε, δίκαιο ανταγωνισμού και αμοιβαιότητα. Ας αναποδηγυρίσουμε λοιπόν τη συζήτηση αυτή βάζοντας την συζήτηση από πάνω προς τα κάτω και όχι ανάποδα. Η ΤΙΖΑ επίσης πρέπει να δώσει μια ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να θέσει τις επιθυμίες, τις ευχές της και ούτω και επομένως και στους κοινωνικούς εταίρους, στους εκπροσώπους της βιομηχανίας, στην κοινωνία των πολιτών γενικότερα και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Πρέπει να είναι ενήμερα τα πρόσωπα αυτά για το τι συζητείτε, ποιος κάνει τι και να δώσουμε την εντύπωση στον κόσμο ότι μπορεί να συνδιαμορφώσει τις διαπραγματεύσεις αυτές. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυξημένη διαφάνεια, βαθιά ριζωμένες αρχές, ένα ρωμαλαίο διάλογο και μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων της Ένωσης και μεταξύ των εταίρων της ΤΙΖΑ και βεβαίως και στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και με το κοινό. Και αυτός είναι και ο σκοπός της ε, παρούσης ε, ε, ακροάσεως. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρέντινγκ για την ξεκάθαρη αυτή τοποθέτηση και για τις πολύ ξεκάθαρες απαιτήσει που εφράσατε. Τώρα, έχουμε το πρώτο πάνελ με όπως είπα μια οριζόντια προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις ΤΙΖΑ. Έχουμε τέσσερις διακεκριμένους εμπειρογνώμονες, τους οποίους θα παρακαλέσω τώρα με τη σειρά να λάβουν το λόγο, να αφαιριστούν σε εννέα λεπτά, για να μας μείνει χρόνος να τους θέσουμε και ερωτήσεις. Πρώτος είναι ο κύριος Ιγνάσιο Διάς, τμήματάρχης στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο κύριε. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να εξηγήσω τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτές τις διαπραγματεύσεις και να εκθέσω κάποια βασικά ζητήματα. Ουσιαστικά θα εκθέσω τους λόγους για τους οποίους διαπραγματευόμαστε. Έχουμε εισέλθει αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, και θα επαναλάβω κάποια στοιχεία που ανέφερε και η κυρία Ρέντινγκ. Ποιο είναι το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης και πώς βλέπουμε τα αμυντικά και επιθετικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα γιατί μετέχει στις διαπραγματεύσεις της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υπηρεσίες και σήμερα είδα ένα πολύ ενδιαφέρον ε, ε, μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για τα, τις υπηρεσίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, αυτό οι υπηρεσίες αντιστοιχούν περίπου στο 70% της οικονομίας μας ε, και έχουμε μεγάλο πλεόνασμα. 150 ε, δις το χρόνο είναι η αξία του πλεονάσματος των υπηρεσιών στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικός είναι ο τομέας και αυτό καλύπτει όλους τους τομείς. Αυτό δείχνει όχι μόνο το άνοιγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ ανοιχτή η αγορά μας για τις ε, υπηρεσίες. Ε, έχουμε και την μελέτη του ΩΣΑ για τους φραγμούς στις χώρες μέλη του ΩΣΑ. Πέραν αυτού, πέρα από αυτό το άνοιγμα, αυτό, μας, ε, αυτό τονώνει και την ανταγωνιστικότητά μας. Αυτό καταδεικνύεται από το πλεόνασμα που έχουμε στο εμπόριο των υπηρεσιών. Παρότι είναι ανοιχτή η αγορά, ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε φραγμούς σε άλλες πιο κλειστές ε, αγορές υπό τη μορφή παραδείγματος χάρη η για τις ισοτιμίες όταν προσπαθεί μια εταιρεία να επενδύσει στο εξωτερικό υπάρχει συνήθως ένα ανώτατο όριο στο ποσοστό που μπορούν να έχουν στα υποκαταστήματά τους σε τρίτες χώρες. Άλλη φραγμή είναι διακριτική μεταχείριση, εξαιρετικά επαχθή διαδικασία διοδότησης, παραδείγματος χάρη. Έχουμε επίσης ε, ρυθμιστικούς ε, φραγμούς, κατ' επίφαση ρυθμιστικούς ε, φραγμούς, αλλά που στόχο έχουν να μην μετέχουν στον ανταγωνισμό δικές μας εταιρείες. Ε, πριν από δύο εβδομάδες ε, είχαμε ένα νέο γύρο των διαπραγματεύσεων και ο τώρα συμμετέχει ε, σε αυτές. Ε, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας ε, είναι ότι ε, δεν θα πρέπει να λειτουργήσει ως εναλλακτική λύση η ΤΙΣΑ σε σχέση με τον ΚΑΤΣ. Αυτή είναι η Συμφωνία των Υπηρεσιών για τον ΠΟΕ. Δεν θέλουμε να έχουμε μια ανταγωνιστική λοιπόν συμφωνία. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ε, μία από τις βασικές, ε, ένας από τους βασικούς όρους ε, που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι πρέπει να επαναλάβουμε τις βασικές παραμέτρους της Συμφωνίας GATS να είναι πανεμφερής η διαδικασία ούτω ώστε να πολυμεροποιήσουμε όπως λέγεται η συμφωνία, τη συμφωνία επιπροσθέτως διαπραγματευόμαστε δηλαδή για την ΤΙΣΑ για να συμβάλλουμε στη συνέχεια στον ΠΟΕ στα πλαίσια της ΓΚΑΤΣ. Δεν ανταγωνιζόμαστε την ΓΚΑΤΣ, θέλουμε να την εξυγχρονίσουμε αυτή τη συμφωνία και θέλουμε μέσω των διαπραγματεύσεων της ΤΙΣΑ να συμβάλλουμε στον εξυγχρονισμό της συμφωνίας ΓΚΑΤΣ. Υπάρχουν άρθρα της ΓΚΑΤΣ που ε, αυτούσια έχουν ε, αντιγραφεί, ε, μεταφερθεί στην ΤΙΣΑ για να είναι πολυμερή η συμφωνία, να αναδειχθεί σε πολυμερή συμφωνία. Τώρα, σας είπα ότι θέλουμε να έχουμε ένα ανοιχτό πνεύμα και όταν έχουμε αυτή την κρίσιμη μάζα θα ε, φέρουμε την τίσα στον ΠΟΗ. Για να επιτύχουμε αυτή την κρίσιμη μάζα θα καλωσορίσουμε νέα μέλη και ε, διαπιστώσαμε ότι για την τίσα στο σημείο 9 το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ε, καλεί τα μέλη να προσπογράψουν τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της ΤΙΣΑ και επιδοκιμάζουμε αυτό το ψήφισμα. Θέλουμε να είναι φιλόδεξη συμφωνία τη. Είναι σημαντικό γι' αυτό. Ο, για ε, η κυρία Ρέντινγκ είπε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού είναι ετερογενή η συμφωνία σε σχέση με το άνοιγμα ως προς το εξωτερικό εμπόριο αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να επιτύχουμε μια νέα ισορροπία και να ε, εισαγάγουμε κάποια στοιχεία αμοιβαιότητας ε, μέσα στη συμφωνία. Φερρυπίν, ε, κάποια πρότυπα για την πρόσβαση στην αγορά, κάποια ε, αυτά που σας είπα για τα ανώτατα όρια για την ισοτιμία, για τις επενδύσεις. Θα υπάρξουν ε, εξαιρέσει, όμω κάποια βασικά στοιχεία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλου του παίκτε τη αγορά πρέπει να κατοχυρωθούν. Α συνοψίσω λοιπόν για ποιο λόγο ε, διαπραγματευόμαστε. Θα ήθελα ε, να ε, καταρρύψω κάποιους μύθους σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες. Δύο είναι τα βασικά στοιχεία. Ποσοτικοί περιορισμοί Πρόσβαση αγορά έτσι ονομάζεται αυτό από τεχνικής πλευράς όταν μιλάμε για διαπραγματεύσεις, δηλαδή από κατά πόσο ανοίγετε την αγορά σας. Επιβάλλεται συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχόντων που πρέπει να είναι υπήκοοι του συγκεκριμένου ε, κράτου για να λάβει επιδότηση ε, μια επιχείρηση. Αυτό σχετίζεται με την ε, πρόσβαση στην αγορά. Και δεύτερον υπάρχει ναι ή όχι διακριτική μεταχείριση. Επιτρέπεται την διακριτική μεταχείριση ανάμεσα στου και και τους ε, ε, αλλοδαπούς παίκτες ε, της αγοράς. Μέσα σε αυτή τη συμφωνία και όλες οι υπόλοιπες συμφωνίες που διαπραγματεύεται για το εμπόριο στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε σαν σχετική ρήτρα. Έχουμε πολύ καλά παραδείγματα γιατί στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ευρύτατο πακέτο μεταρρυθμίσεων στο πακέτο για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μετά την κρίση που σημειώθηκε στην Ευρώπη και έχουμε εξαιρετικά εκτεταμένες δεσμεύσεις και στην ΚΑΤΣΕ e και σε άλλες συμφωνίες σε Ελευθέρου Εμπορίου FTAs. Λοιπόν, έχουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και αυτό έχει γίνει με, κατάργηση της διακριτικής μεταχείρισης. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός μέσα από τους ποσοτικούς περιορισμούς που έχουμε επιβάλει. Δεν περιορίζουμε Δεν έχουμε επιβάλει αυτούς, ε, τις, ε, αυτούς περιορισμούς ε, και από την άλλη δεν περιορίζουμε το πεδίο των διαπραγματεύσεων μέσω των ποσοτικών περιορισμών. Στη συνέχεια έχουμε οριζόντια αλλά και τομεακά κεφάλαια για την εγχώρια νομοθεσία, για τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες αδειοδότησης ουσιαστικά. Περί αυτού πρόκειται και συζητούμε ζητήματα οικονομικής διακυβέρνησης όταν οι νομοθέτες για τις τηλεπικοινωνίες δεν πρέπει να έχουν σχέση με τους παρόχους ε, όταν ε, επίσης ε, εξετάζουμε το θέμα της απλούστευσης της διαδικασίας αδειοδότησης για τους φορείς αγοράς στις τηλεπικοινωνίες. Λοιπόν, αυτά για το για τις διαπραγματεύσεις ας περάσουμε στα επιθετικά και αμυντικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδόν σε όλους τους τομείς έχουμε πλεόνασμα και είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για τις τηλεπικοινωνίες, για τις επαγγελματικέ υπηρεσίες, για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με υπολογιστές. Έχουμε επιθετικό συμφέρον λοιπόν. Ε, για τις δημόσιες προμήθειες ε, έχουμε καταθέσει πρόταση για έξι σημεία για κατάρριξη διακριτικής μεταχείρισης για τους δικούς μας φορείς. Λέμε στα ε, ε, υπόλοιπα συμβαλόμενα μέρη ότι δεν θα πρέπει ε, να υπάρξει κατα... διακριτική μεταχείριση ως προς τους φορείς μας που δραστηριοποιούνται στις χώρες σας. Αυτό είναι βασική απέτηση που έχουμε από την ΤΙΣΑ. Κλείνοντας, όπως είπε και η κυρία Ρέντινγκ, υπάρχουν τομείς όπου δεν είμαστε ε, αμυντικοί επειδή δεν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά δεν θέλουμε να αναλυθούν δεσμεύσει που δεν μπορούν να εκπληρωθούν. Οι υπηρεσίε όπου, παραδείγματο χάρη, ακολουθούμε την πάγια γραμμή μα από την ΓΚΑΤΣ και μετά και που έχουμε διατηρήσει όλε τι FTA που έχουμε διαπραγματευτεί ε, μέχρι στιγμή σε μονοπόλια και αποκλειστικά δικαιώματα σε όλε τι δημόσιε υπηρεσίε που ε, καλύπτουν υπηρεσίες σε όλους τους τομείς ε, και αποκλείεται δέσμευση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση για την δημόσια υγεία, για την παιδεία, για τα οπτικοακουστικά ή για την ε, υδροδότηση, την ίδρυυση. Ε, θα θέλουμε λοιπόν να κατοχυρωθεί η θέση μας σε αυτό το κύριο σημασία σημείο. Άλλη, άλλα μέλη θα ε, προτείνουν ε, ίσως άλλα, άλλους τομείς ε, πέραν του εμπορίου, παραδείγματος χάρη ασφάλειες, υγεία. Μα ήρθε μια πρόταση πριν από δύο εβδομάδε. Ήταν ξεκάθαρη αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε, σε καμία περίπτωση δεν θα συμφωνήσουμε σε μια πρόταση που σχετίζεται με την κινητικότητα στον τομέα των υπηρεσιών υγείας. Θα σταματήσω εδώ γιατί δεν έχω χρόνο. Σας ευχαριστούμε λέει ο κύριος Λάγκε. Ήδη σας ήταν πληρέστατος. Ο καθηγητής ε, Δ. Μάρκους Κραγέσκη, καθηγητής ε, Δημοσίου και Διεθνούς Δικαίου από το Πανεπιστήμιο Ερλάνγκεν Νιρεμβέργης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση με χαρά και τιμή είμαι εδώ να σας μιλήσω. Θα αναφερθώ σύντομα σε κάποια σημεία. Καταρχάς να πω και είναι σημαντικό ότι παρόλο που είχαμε 10 γύρους διαπραγματεύσεων δεν είναι και τόσο γνωστά αυτά. Έχουν δημοσιευτεί βεβαίω κάποια στοιχεία για τους γύρους διαπραγματεύσεων αλλά το σημαντικό είναι οι συγκεκριμένε προτάσεις που υπάρχουν. Αναφέραμε με για την Τουρκία, ας πούμε. Σχετίζονται και με τις υπόλοιπες προτάσεις αυτές. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι συνδέεται με αυτές τις διαπραγματεύσεις και δεν ξέρουμε και τι αιτήματα υπάρχουν από τους συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις αυτές. Συνεχίζουμε λοιπόν να εικάζουμε για το στόχο αυτών των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να μιλήσω για τρία σημεία. Το γενικό πλαίσιο και την δομή αναφέρθηκε ήδη. Βεβαίως ο περίνας εδώ βασίζεται στο GATS. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά σε σχέση με το GATS, δηλαδή η προσέγγιση σε σχέση με τις δεσμεύσεις. Μια ευρυδική προσέγγιση ακολουθεί η ΤΙΣΑ ένα κατάλογο δηλαδή θετικών και αρνητικών στοιχείων. Δύο κυρία ερωτήματα έχουμε εδώ. Τι καλύπτει η αρνητική λίστα και τα στοιχεία της, οι υποχρεώσεις οι εθνικές ενδεχομένως, αλλά και άλλα μπορεί στοιχεία. Θέματα που αφορούν διαφάνεια και τις διαφορές χώρες, αλλά και θέματα πρόσβαση στις αγορές. Αν κατάλαβα καλά και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, υπάρχουν θέματα που αφορούν την πρόσβαση στις αγορές και τα πλαφόν. Στο παρελθόν είχαμε μια οριζόντια προσέγγιση στις εμπορικές συμφωνίες και αυτά τα στοιχεία πρόσβασης αγοράς ήταν στο αρνητικό κατάλογο. Έτσι Μειώναμε βεβαίω και το πεδίο των... τη θετική λίστα, του δικού καταλόγου. Αν κατάλαβα πάντω καλά την πρόταση από το κείμενο, εδώ στους ορισμούς υιοθετούμε κάτι το οποίο μοιάζει με το παράρτημα 2 και το σύστημα εκεί. Γιατί μιλάει για τωρινά και μελλοντικά μέτρα. Όμως οι ίδιες διατάξεις περιλαμβάνουν αυτό που λέμε μηχανισμό του παραρτήματος 1. Και δεν είμαι καθόλου βεβαίως το πώς αυτά συνδυάζονται. Εμένα μου φαίνεται τουλάχιστον ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια εδώ για να δούμε ακριβώς πώς αυτή η υβριδική προσέγγιση εφαρμόζεται, αν συνδυάσουμε δηλαδή την προσέγγιση αρνητικής και θετικής λίστας. Υπάρχουν και δυσκολίες βέβαια που θα ήθελα να αναφέρω Δηλαδή με τη χρήση αυτής της μοναδικής προσέγγισης είναι σχετικά δύσκολο για τους εμπλεκόμενους αλλά και για τους ρυθμιστές και τους ευρωβουλευτές να συγκρίνουν τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η Ένωση μέχρι τώρα εκτός από την ε, Συμφωνία ΣΥΤΑ που ήταν ε, βασισμένη σε μια θετική λίστα, σε ένα θετικό κατάλογο αλλά δεν ξέρουμε τι περαιτέρω δεσμεύσει θα αναλυφθούν και πόσος καιρός θα χρειαστεί. Θα ήθελα επίσης να πω ότι όχι μόνο οι ρυθμιστές, η ΜΚΟ και το κοινό, αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έπρεπε να ωφεληθούν από αυτές τις δεσμεύσεις. Το θέμα λοιπόν παραμένει κατά πόσο κατανοούν την διάρθρωση, την δομή αυτών των δεσμεύσεων και αυτό θα ήθελα να το υπογραμμίσω. Δεύτερο σημείο αφορά τις εθνικές νομοθεσίες. Αναφέρθηκε και στις εμπορικές επαφές όταν μιλάμε για τις εθνικές νομοθεσίες και κανονισμούς μιλάμε για ένα horizontal necessity test και για το ΣΥΤΑ βλέπω ότι ο κανονισμός δεν περιλαμβάνει αυτή την δοκιμασία ανάγκης οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί κανείς να διαφωνήσει, οπότε μπορεί να πάρει ως μοντέλο το κείμενο της ΣΥΤΑ. Και άλλοι εταίροι, ιδιαίτερα αυτή τη ΣΤΙΖΑ, συμφωνούν με αυτή τη δοκιμασία, οπότε πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Επίσης, έχουμε έγγραφα τομέκης, αναφοράς ή συγκεκριμένα ρυθμιστικά τομεακά σχέδια όπως ας πούμε στις τηλεπικοινωνίες στα πλαίσια του ΓΚΑΤ αλλά έχουμε και άλλες προτάσεις για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ας πούμε υπάρχουν προτάσεις και για το τομέα της υγείας σημαντικά όλα αυτά και θα ήθελα να πω ότι από ό,τι καταλαβαίνω εγώ την πρόταση αυτό ακόμα δεν έχει συζητηθεί στα πλαίσια του εμπορίου παρόλο που βεβαίως υπάρχουν δεσμεύσεις γκάτς από άλλε χώρες και υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά το κατά πόσο μπορείς να μεταφέρεις την ασφάλεια. Υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί και είμαι βέβαιος ότι αν είναι τη γνώμη κάποιο ότι αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει τμήμα των διαπραγματεύσεων, τότε μπορούμε να το ακολουθήσουμε ω θέση. Όμως, εγώ θα έλεγα ότι αυτό δεν βρίσκεται τελείως εκτός μιας ατζέντα εμπορικής υπό ευρία έννοια. Τέλος, κοινοφελείς υπηρεσίε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι στις προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες της Ένωσης είχαμε διάφορα εργαλεία και μηχανισμούς για να πετύχουμε αυτό που είπε η κυρία Ρέντινγκ, δηλαδή να διατηρήσουμε εκτός της κοινοφιλής υπηρεσίες. Όμως, αν δούμε αυτά τα εργαλεία πιο προσεκτικά, θα δούμε ότι δεν υπάρχει οριζόντια οριζόντιος αποκλεισμό ή εξαίρεση των κοινωνικών των δημοσίων υπηρεσιών. Έχουμε μόνο κάποια παραδείγματα που αφορούν κυβερνητικές αρχές. Θα ήθελα να πω μόνο ότι αν δούμε την ιστορία των διαπραγματεύσεων των εμπορικών, πριν από 15 χρόνια είχαμε μεγάλες συζητήσεις για τις κοινοφιλείς υπηρεσίες και τον ΚΑΤΣ και πολύ ακριβώς επιχειρηματολόγησαν ότι αυτή ακριβώς η εξαίρεση των κοινοφιλών υπηρεσιών θα τις προστατεύσει αλλά κανείς δεν το λέει πια σήμερα αυτό. Λέμε σήμερα ότι οι κοινοφελείς ταυτίζονται με τις ε, υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα και θα πρέπει να εξαιρεθούν. Αλλά πρέπει να δούμε και πάλι ποιος είναι ο ορισμός, ε, τι θα εξαιρεθεί κτλ. Εξάλλου έχουμε και κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις στα πλαίσια συμφωνίας με τη Σιγκαπούρη. Αλλά βεβαίως η ρήτρα για τις κοινοφελείς επιχειρήσεις νομίζω αποκλεί μόνο τα μονοπόλια και τους παρόχους υπηρεσιών. Οπότε οποιοδήποτε άλλο εργαλείο δεν εξελείται, οποιοδήποτε άλλο εργαλείο δεν εξελείται από αυτή την ρήτρα. Επίσης, μια σημαντική προσθήκη στην εργαλειοθήκη είναι ο ορισμός αυτών των υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από, δημόσιο, από δημόσια κονδύλια. Θεωρώ ότι είναι αρκετά ευρεία ως ε, ορισμός η αναφορά αυτή. Και νομίζω ότι αυτό είναι θετικό, αποτελεί ένα επίτευγμα και νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει κάλλιστα τμήμα των διαπραγματεύσεων ΤΙΖΑ ή και το δεσμεύσεων στα πλαίσια του TTIP. Ένα τελευταίο σημείο να υπογραμμίσω, οι εξαιρέσεις για τοπικά μέτρα. Η κυρία Ρέντινγκ αναφέρθηκε στις γενικές αρχές που θα πρέπει να μας καθοδηγούν το πρωτόκολλο 26 που ιδιαίτερα αναφέρεται στη διακριτική ευχέρεια των αρχών να παράσχουν αυτές τις υπηρεσίες στους άμεσους καταναλωτές, δηλαδή τοπικές αρχές κτλ. Και πάλι εδώ νομίζω είναι σημαντικό να δούμε ακριβώς και να εξετάσουμε αυτά τα τοπικά μέτρα και να διατηρήσουμε τα υπάρχοντα μέτρα, κάτι το οποίο δηλαδή ήδη έχει επιτευχθεί στα πλαίσια του ΣΥΤΑ, αλλά να διαφυλάξουμε και το μέλλον των τοπικών μέτρων. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η παραπομπή στα τοπικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1, αλλά στο παράρτημα 2. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για αυτή την πολύ ενημερωτική εισήγηση Επόμενος ομιλητής, η κυρία Πένι Κλάρκ, Γενικός Γραμματέας της, ε, στην υπηρεσία για τις δημόσιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Θα αρχίσω ίσως ε, ε, με κάτι που είπατε εσείς κύριε Λάγκε. Δύο επάναλ έχουμε, το οριζόντιο και το τομεακό. Ε, αλλά για τον τομέα της υγείας ε, μας ενδιαφέρουν και τα δύο, διότι ο στόχος ε, είναι και τομεακός και οριζόντιος στον τομέα της υγείας. Θα πρέπει αυτό να ενσωματωθεί σε μια σειρά από πολιτικές, όχι μόνο στη πολιτική στον τομέα της υγείας, εξού και η σχέση με τον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών. Εγώ σε αυτό θα επικεντρωθώ. Θα ήθελα επίσης να πω πως έχουμε διάφορες ανησυχείς για άλλα οριζόντια ζητήματα, μεταξύ των οποίων οι συνθήκες εργασίας, ε, δικαιώματα, συνδικαλιστικά, ε, ε, ισότιμη μεταχείριση εργαζομένων και ούτω καθεξής. Νομίζω κάποια, κάποια άλλη στιγμή μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτά. Τέλος πάντων, όταν μιλούμε για τις υπηρεσίες, και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στην σημασία των υπηρεσιών, όπως και η κυρία Ρέντινγκ, ε, εκφύσεως ε, ε, οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν στενότερη σχέση με το, την εγχώρια κατάσταση σε σχέση με τις υπηρεσίες, σχετίζονται με τους ανθρώπους, δηλαδή η ποιότητα των υπηρεσιών συνδέεται άμεσα με την, τους παρόχους. Για την ετυποποίηση πρέπει οπωσδήποτε να περάσουμε από κατοχήρωση των εργασιακών δικαιωμάτων, καταλαβαίνετε. αλλά ξαναλέω, έχουν πιο τοπικό υφή σε σχέση με τις υπηρεσίες και η έλλειψη ανταγωνισμού δεν συνεπάγεται άμεσα ότι υπάρχουν φραγμοί, ε, όπως είπαν οι συνάδελφοι για το εμπόριο των υπηρεσιών. Δεν θα πρέπει δηλαδή να υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει διασυνοριακό εμπόριο και άρα αυτό σημαίνει αυτόματο ότι υπάρχουν ακόμη φραγμοί. Θέλουμε ρήτρες διασφάλισης για τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως σωστά αναφέρθηκε, διότι αυτό σχετίζεται με τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις δημόσιες υπηρεσίες και βλέπουμε λοιπόν ότι ε, ε, αυτό που επιδιώκουμε είναι προς τα πάνω να ε, ευθυγραμμιστούν οι κοινωνίες της Ευρώπης για την υγεία, για την ποιοτική παιδεία, για το καθολικό δικαίωμα, οικουμενικό δικαίωμα πρόσβασης στο νερό που έχει κατοχυρωθεί από τον ΟΗΕ. Θέλουμε να προωθήσουμε την απασχόληση, την ανάπτυξη, διότι η επένδυση που γίνεται από το κράτο στι δημόσιε υπηρεσίες έχει τέτοια αποτελέσματα και πάντοτε θα πρέπει να γίνονται όλα αυτά προς συμφέρον των πολιτών που χρειάζονται αυτέ τι υπηρεσίε. Άρα θα πρέπει θετικά να προσεγγίσουμε το ζήτημα. Τι συμβλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και θα πάρω το θέμα τη υγειονομική περίθαλψης γιατί είναι ε, στα πλαίσια τη συζήτησή μα ένα πολύ βασικό σημείο σε σχέση με το τι θέλουμε για το μέλλον και ποιε διαρροέ υπάρχουν προ τα έγγραφα. Λοιπόν, βλέπουμε την αρμοδιότητα και όταν συζητούσα με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα ή στη Λετωνία παραδείγματο χάρη για την έλλειψη πρόσβασης ε, στις υπηρεσίες υγείας ε, και λέμε ότι είναι οικουμενικό δικαίωμα και κατοχυρώνεται τη κάτω θυμολογιών δικαιωμάτων ε, ενέκρινε μια ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου καλεί για έγκριση μέτρων βάσει προσέγγιση checklist για τα βασικά δικαιώματα. Βλέπουμε λοιπόν κάποιοι συνάδελφοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λένε ναι, ναι, ναι, αλλά δείτε και τι κάναμε με την κινητικότητα στον τομέα της υγείας. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τα συστήματα ε, προστασίας, ε, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη γάμα δέλτα απασχόλησης. Αν θέλετε όμως να το προσεγγίσετε από πλευράς ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, τότε είναι μάλλον αρμοδιότητα της γάμα δέλτα δικαιοσύνης. Αν θέλετε να δείτε τις σχέσεις με την οικονομική διακυβέρνηση, θα πρέπει να αποταθείτε στην έκφυνη. και υπάρχουν συστάσεις που ε, σχετίζονται με αυτού του διαφορετικού τομεί, Ο απότερο στόχο, η προώθηση καλής, ε, καλών υπηρεσιών υγεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, Α, και ξέχασα ότι υπάρχει και αυτό το θέμα τη σύγκρουση των αρμοδιοτήτων ε, που επηρεάζει επίσης την έκβαση του παιχνιδιού, διότι θέλουν τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο να νομοθετούν και να ρυθμίζουν τις δημόσιε υπηρεσίε. Είναι μεικτή η αρμοδιότητα λοιπόν, οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για απελευθέρωση, διότι αναφερθήκαμε και στο Συμβούλιο και είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο του σε αυτό το τομέα. Έχει εγκρίνει πάρα πολύ καλέ αρχέ σε σχέση με την ε, περίθαλψη ε, που πρέπει να εφαρμοστούν. Αυτός είναι ο ρόλος των δημοσίων υπηρεσιών, πώς κατοχυρώνεται, ε, πώς η TSA και η TTIP επηρεάζουν τις δημόσιες υπηρεσίες. Είναι ένα πλέγμα για μας. Ό,τι βαραληφθεί σε μια συμφωνία μπορεί να συμπεριληφθεί σε μια άλλη ε, και όπως είπατε έχει ήδη εγκριθεί, υιοθετηθεί η ΣΥΤΑ ε, και ε, πραγματικά πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει τη ΣΥΤΑ διότι είναι μια, ένα κρατέο έρισμα για μας. Ξέρουμε τι μπορούμε επιπλέον να συμπεριλάβουμε σε μια νέα συμφωνία. για τις δημόσιες υπηρεσίες και τον αποκλεισμό τους από τις διαπραγματεύσεις. Ο συνάδελφος δίπλα είπε ότι ε, προς το παρόν δεν έχουν αποκλειστεί οι δημόσιες υπηρεσίες σε καμία από τις εμπορικές ε, συμφωνίες. Όμως ακούγοντας τον υπόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνω πως ε, υπάρχει μια βούληση να υπάρξει κατανόηση ότι πρέπει να προστατεύσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες για την πρόσβαση στην αγορά και ε, φυσικά έχουν γίνει βήματα, αλλά έχουμε ακόμη ανησυχίες ε, διότι δεν εξυπηρετούνται πλήρως ε, οι στόχοι μας να έχουμε μια οικουμενική πρόσβαση στην υγεία, μάλλον καθολική πρόσβαση στην υγεία σε όλα τα κράτη-μέλη και δεν είμαι σίγουρη αν εξυπηρετείτε το δημόσιο συμφέρον ναι, με την προσέγγιση που έχετε υιοθετήσει, αλλά ξεκάθαρα υπάρχει μια βούληση. Λοιπόν, στην ΤΙΖΑ, όπως είπατε, <clears throat> κυρία Ρέντινγκ, η ΤΙΖΑ είναι ε, μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες. Γιατί να μην είναι αυτή η πρώτη συμφωνία όπου, πραγματικά θα αποκλειστούν από τις διαπραγματεύσεις ε, και θα προβλεφθούν οι σχετικές ε, διατάξεις για τις δημόσιες υπηρεσίες για την κατοχυρωσή τους. Για τα τεχνικά ε, σημεία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμπεριληφθούν στις διαπραγματεύσεις ε, όταν αλλάζουμε με την υβριδική προσέγγιση και περνάμε ε, από, τον αρνητικό στο θετικό κατάλογο δυσκολεύομαι και εγώ η ίδια να καταλάβω περί ως πρόκειται οπότε φανταστείτε οι άλλοι ε, και θα πρέπει να προσέξουμε διότι διαρκώς γίνονται αλλαγές και ο Μάρκους είπε ότι αυτή η αλλαγή από, την, ε, τον αρνητικό στο θετικό κατάλογο, την ευρυδική προσέγγιση, Δηλαδή ό,τι είναι στο θετικό κατάλογο δεν είναι στον αρνητικό και άρα δεν είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ε, σκέφτομαι, ωραία, πώς θα τα κατανοήσουν ε, αυτοί που διαπραγματεύονται αυτά. Ο στόχος είναι να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και ε, ανάπτυξη των ενδογενών ικανοτήτων κατανόησης ε, και επ' αυτού νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει και να συμβάλλει ούτως ώστε να καταλάβουμε όχι τι σημαίνουν αυτές, αυτοί οι όροι, αλλά ποιος είναι ο στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο και των υπολείπων ε, μέρων που διαπραγματεύονται, διαφυλάττοντας ε, τις αξίες ε, και τις αρχές μας, ε, στην προόδο αγωγή ενός, ε, ε, μιας κοινωνικής διάστασης του εμπορίου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και σε αυτό το τομέα, στο κοινωνικό τομέα, ε, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο το εμπόριο. Σχεδόν έχω ολοκληρώσει. Ήθελα μόνο να σχολιάσω κάποια ειδικότερα σημεία για τα υπέρ και τα κατά της ΤΙΖΑ. Ε, ε, περιμένουμε ακόμη την ε, αξιολόγηση αντικτύπου, βιώσιμο ε, βιώσιμου αντικτύπου. <coughs> Ε, διότι νομίζω δεν έχουμε δει ποια είναι τα θετικά στοιχεία ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι για την υγεία ένα ε, παράδειγμα που χρησιμοποιούμε με τους συναδέλφους και στο Κοινοβούλιο είναι η ιδέα μιας νέας δημόσιας υπηρεσίας. Δεν περιοριζόμαστε στο να διαφυλάξουμε τα κεκτημένα, ε, επιδιώκουμε και νέους στόχους στη μακροπρόθεσμη υγειονομική περίθαλψη και στην προστασία στην Επιτροπή Κοινωνική Προστασία έχουν ήδη συμφωνήσει η Επιτροπή και το Συμβουλίο για μια σειρά συστάσεων. Η πρώτη είναι ισοτιμία, αποτελεσματικότητα, ήθο σε σχέση με την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων κινδύνων και την ενσωμάτωσή του στο σύστημα κοινωνική ασφαλή, αμοιβαιοποίηση, αν θέλετε, των κινδύνων. Δεν ε, ε, επιθυμούμε αποκλεισμού λοιπόν σε αυτό το τομέα. Αντίθετα, αναρωτιόμαστε πω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός μπορούμε ε, μακρόπνοα να αναπτύξουμε ένα βιώσιμο σύστημα υγεία και περίθαλψης. Ευχαριστούμε. τελευταίο ομιλητής, ο κύριος Πασκάλ κερνή, που είναι εκτελεστικός διευθυντής στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Υπηρεσιών. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση κύριε Πρόεδρε να συμμετάσχω στο πάνελ. Η οργάνωσή μου εργάζεται ιδίω στο εμπόριο, αποκλειστικά στο εμπόριο υπηρεσιών και αυτό είναι σημαντικό. Πρώτα, για τις διάφορες προσφορές πρόσβαση στην αγορά. Ευχαριστώ βέβαια την εισηγήτρια κυρία Ρέντινγκ πρώτα που έβαλε σε αυτές τις ε, πέντε κιανές γραμμές και τις πέντε ερυθρές γραμμές. Για την ίδια τη δομή τώρα, αυτή η υβριδική προσέγγιση μας φαίνεται λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί. Εμείς έχουμε αρνητικό κατάλογο που είναι απλούστερος να κατανοηθεί από τις εταιρείε αλλά και από τον καθένα δηλαδή τελικά. Βέβαια θα θέλαμε να επεκταθεί η συμφωνία και σε άλλες χώρες και γι' αυτό εάν κάποιες χώρες προτιμούν το θετικό κατάλογο αυτό είναι ένα σημαντικός λόγος. Και βεβαίω να προσπαθήσουμε να δώσουμε πολυμερή χαρακτήρα στην ε, συμφωνία. Να παραμείνει η δομή GATS στην ΤΙΣΑ, να μην αρχίσουμε δηλαδή από το μηδέν. Υποστηρίζω επίσης την ιδέα να χρησιμοποιήσουμε κάποια, κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές, όλες οι χώρες δηλαδή, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε ταχύτερα σε μια απελευθέρωση για τις χώρες. Να δούμε τις διάφορες χώρες. Είναι 24 χώρες γύρω από το τραπέζι. Με πολλές από τις χώρες αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη διαθέτει συμφωνίες είτε ήδη υπογεγραμμένες είτε υποδιαπραγμάτευση. Θα θέλαμε λοιπόν η ΤΙΣΑ να στοχεύσει στις χώρες εκείνες όπου δεν έχει συμφωνίες πρόσβαση στην αγορά η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζω εδώ με κόκκινο Αυστραλία, Χονγκ Ισραήλ, Ταϊβάν, Νέα Ζηλανδία, Πακιστάν, Παραγουάη, Ουρουάη και την Τουρκία. Και την Τουρκία. Ιδιαίτερα δε για την Τουρκία που είναι και η γειτονική μας χώρα. Μεγάλη χώρα με σημαντική ανάπτυξη. Δεν έχουμε στο σύμφωνο ακόμα με την Τουρκία. Έχουμε τελωνιακή μεν ένωση, δεν έχουμε όμως συμφωνία για τις υπηρεσίες εκτός από την δέσμευση Γκάτς που δεν είναι και πολύ υψηλό επίπεδο για την θέσπιση κανόνων στην ΤΙΣΑ. Το υποστηρίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγησε ποια πράγματα έχουν τεθεί επιτάπητος ήδη. Η κατάργηση των licensing procedures που είναι περίπλοκες, αλλά τουλάχιστον να υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις που να είναι ε, να επιβάλλουν μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτό ζητούν όλες οι χώρες για την προσωρινή κινητικότητα του προσωπικού. Επίσης εδώ μιλήσαμε για τηλεπικοινωνίες, για ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Επίσης, όταν θα μπουν στις ρυθμίσεις αυτές και οι κρατικές επιχειρήσεις. Ζητούμε και εκεί να υπάρξει και ε, πρόσβαση στην αγορά. Να δούμε τώρα τις πέντε ε, και γραμμές που εξέτασε η συγκεκριμένη και τις έθεσε υπόψη μας και αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Να δούμε ποια είναι η θέση μας επ' αυτού. Η ανάγκη αμοιβαιότητας. Βεβαίως κατανοούμε ως αμοιβαιότητα κάτι ευρύ, δηλαδή όλες οι χώρες να ανοίξουν λίγο πολύ, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι όμως σε κάθε μεμονωμένο τομέα. Αν δηλαδή στον τάδε τομέα έχει ανοίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει και η άλλη χώρα. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Δεν είναι και το πνεύμα άλλωστε που μας ενδιαφέρει. Θα θέλαμε βέβαια όλες οι χώρες να ανοίξουν περισσότερο. Ένας από τους λόγους για τους οποίους υπάρχει η ΤΙΖΑ είναι διότι η DDA δεν προχωρεί καθόλου. Και εμείς του τομέα των, ε, των ε, υπηρεσιών ε, αισθανόμαστε όμοιροι της γεωργίας. Θέλουμε να προχωρήσουν λοιπόν όλες οι χώρες τώρα. Για την δεύτερη και τρίτη και ανή γραμμή, ε, για τις διεθνείς προδιαγραφές των υπηρεσιών και για να προσφερθούν συγκεκριμένα απτά ωφελήματα στους ε, Ευρωπαίους πολίτες, ασφαλώς τις υποστηρίζουμε τις γραμμές αυτές. Εκτός από αυτές, θέλουμε η ΤΙΣΑ να υποστηρίξει και να δημιουργήσει νέες προδιαγραφές, νέα στάνταρτ να μπουν λοιπόν προδιαγραφές στην ΤΙΣΑ ώστε όλες οι ανεπτυγμένες χώρες να βάλουν κοινέ προδιαγραφές στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Εκτός από τους τομείς που αναφέραμε προηγουμένως έχουμε επιθετικά εντό εισαγωγικών ε, ενδιαφέροντα και σε άλλους τομείς και σε υπηρεσίες. Για παράδειγμα στην εφοδιαστική και σε νέες υπηρεσίες που αναπτύσσονται τώρα ταχύτατα όπως περιβαλλοντικές ή σε σχέση με την ενέργεια όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, σημαντική ικανότητα ανάπτυξης. Έρχομαι στην Κίνα. Βέβαια και θέλουμε η Κίνα να μπει στο παιχνίδι, on board δηλαδή, γιατί θέλουμε η ΤΙΣΑ να επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Και οι χώρες BRICS και ASEAN για παράδειγμα επίσης μας ε, φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον και το υποστηρίζουμε. Έχουμε ταχθεί άλλωστε υπέρ της συμμετοχής στην ΤΙΣΑ της Κίνας. Η Κίνα ήδη έχει εγκρίνει και προχωρεί σε κάποια σε βάθος μεταρρύθμιση για τις επενδύσεις και ανοίγει επίσης και ζώνες ελεύθερων συναλλαγών όπου ε, μπορούν να ε, υπάρξει ανταλλαγή υπηρεσιών. Ακούσαμε όμως πρόσφατα και ένα project για κυβερνοασφάλεια που θα αναπτυχθεί όπου η Κίνα πρόκειται εκεί ωστόσο να ορθώσει νέους φραγμούς. Αυτό για μας είναι σημαντική απειλή και διορωτώμεθα αν εδώ η Κίνα κάνει κάποιο παιχνίδι. Δηλαδή θέλουμε να μπει η Κίνα μέσα, αλλά όχι να κλείσει περισσότερο, να ανοιχτεί περισσότερο. Η Ουρουγουάη μπήκε προ δύο εβδομάδων νομίζω. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι η αντίδραση της Κίνας. Θα παραμείνει ήρεμη ή θα πει ξαφνικά «Α, δεν θέλω τώρα πια να μπω στην Τίσα». Αυτό είναι το μέγα ερωτηματικό. Εμείς φοβούμεθα την αδυναμία να επεκταθεί η Τίσα. Είπαμε θέλουμε η Τίσα να προχωρήσει. 24 χώρε δεν φτάνουν. Η τελευταία η γραμμή λοιπόν, υποχρέωση, ε, μάλλον δέσμευση της ΤΙΣΑ να εφαρμοστεί και γιατί όχι να έχουμε τον μηχανισμό ε, ρύθμισης διαφορών του ΠΟΕ. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό, διότι πολλές χώρες του ΠΟΕ δεν υποστηρίζουν ακόμα τουλάχιστον την ΤΙΣΑ και μπορεί να πούν όχι, διότι οι κανόνες για να υιοθετηθεί το ε, σύστημα του ε, ΠΟΕ θα είναι όλες οι χώρες να παραχωρήσουν αυτή την εξαίρεση του waiver. Και χρειαζόμαστε λοιπόν ιδιαίτερο μηχανισμό ε, επίλυση των διαφορών στην ΤΙΣΑ. Πέρσι, ωστόσο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε κανονισμό που λέει καθαρά ότι δεν μπορείτε να προβαίνετε σε αντίπεινα στον τομέα των υπηρεσιών. Θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εφαρμοστεί η ΤΙΣΑ. Οι πέντε ερυθές γραμμές τώρα υπηρεσίες καθολικού ενδιαφέροντος και ε, κοινοφελείς υπηρεσίες. Αυτό το υποστηρίζουμε. Δεν θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων στην ΤΙΣΑ. Εκεί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια προστασία για τις υπηρεσίες αυτές και η οποία πρέπει να ενισχυθεί και γιατί όχι. Το κεφάλαιο περί κινητικότητας τώρα. Εδώ μου φαίνεται να υπάρχει κάποια σύγχυση. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει δεσμεύσει για την προσωρινή κινητικότητα των επιχειρηματιών. Περί αυτού πρόκειται εδώ. Εμεί θέλουμε μάλιστα περισσότερο, εντονότερα το στοιχείο αυτό μέσα στην ΤΙΖΑ. Δεν μιλούμε για μετανάστευση, δεν μιλούμε για χορήγηση προξενικών θεωρήσεων, δεν μιλούμε για αυτά τα πράγματα. Μιλούμε να ανοίξει η προσωρινή κινητικότητα των επιχειρηματιών και θέλουμε ΤΙΖΑ να το ανοίξει αυτό περισσότερο. Το δικαίωμα ρύθμισης. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε γιατί. Βέβαια κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να ρυθμίζει. Δεν υπάρχει καμία διεθνή συμφωνία που μπορεί να ε, απαγορεύσει κάποια χώρα να προβαίνει σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Βέβαια η χώρα μέλος θα διατηρεί το δικαίωμα να ρυθμίζει, ωστόσο με συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Για το κοινωνικό ντάμπινγκ για μας είναι το ίδιο βλέπουμε ότι υπάρχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν αμφισβητείται το ε, κοινοτικό κεκτημένο. Η τελευταία ερυθρά γραμμή, η τελευταία κόκκινη γραμμή είναι η προστασία των δεδομένων. Εμείς στην ESF έχουμε ασχοληθεί πολύ εντατικά με αυτό. Καταλήξαμε σε ένα συμβασμό και είπαμε και βέβαια η ρύθμιση προστασίας δεδομένων δεν πρέπει να αμφισβητείται από μια εμπορική συμφωνία. Όμω η εμπορική συμφωνία είναι και μεγάλη ευκαιρία για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα ηγερθούν νέοι φραγμοί για την μεταφορά δεδομένων. Μεταφορά δεδομένων είναι στην ουσία παροχή εμπορικών υπηρεσιών. Δεν υπάρχει καμία εμπορική υπηρεσία στον κόσμο χωρί μεταφορά δεδομένων. Αυτό πρέπει να τονιστεί σαφέστατα και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, μεν προστασία δεδομένων, αλλά και θέσπιση κανόνων που θα επιτρέπουν την μεταφορά δεδομένων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν τοπικέ ρυθμίσει που να κάνουν τη ζωή μα πιο δύσκολη. Αυτά, ευχαριστώ. Τώρα λαμβάνουν το λόγο τα μέλη, Εσεί πρώτοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που είπε η κυρία Ρέντινγκ στην αρχή. Δηλαδή, κυρίως για την έναρξη μιας δημόσιας συζήτησης για αυτά τα θέματα και για την ύπαρξη, ανάγκη ύπαρξης διαφανούς δημόσιας συζήτησης για τη ΤΙΖΑ ενώ των διαπραγματεύσεων. Αν δεν γίνει αυτό, θα καταλήξουμε σε συζητήσεις που θα περιπλέξουν τα πράγματα, θα δημιουργήσουν σύγχυση. Αν θυμάστε μετά την ΓΚΑΤ είχαμε την συζήτηση για την ΑΚΤΑ. Οπότε η ΤΙΣΑ αν δεν ακολουθήσει αυτή η πορεία θα γίνει μια πολύ δύσκολη υπόθεση στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να πιέζουμε για μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με το τι ακριβώς βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Και μιας και διαπραγματεύονται όλα αυτά μαζί με τον ΠΟΕ, εμείς πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση σύμφωνα με τους κανόνες διαφάνειας του ΠΟΕ. Και αυτό που προγουμένος, ο Μάρκος προηγουμένως, δηλαδή οι προσφορές και από τις δύο πλευρές πρέπει να είναι δημόσιες ώστε να μπορούν να εξεταστούν για την διαφάνεια. Τι κάνει η Κομισιόν ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Η εντολή είναι μεγάλο βήμα, αλλά θα είναι κενό περιεχομένο αν δεν συνοδεύεται από τίποτα άλλο. Δεύτερη ερώτηση. Γκάτς. Αφορά και τον Μάρκος αυτή η ερώτηση. Στο Γκάτς υπάρχει η δυνατότητα τα μέρη να αποσυρθούν, μάλλον να αποσύρουν υπηρεσίες και τομείς από τις προσφορές τους. Τι γίνεται με τους αντίστοιχους κανόνες για την ΤΙΖΑ. Εντάξει, πολύ ωραία. Όταν περιλαμβάνεται κάτι και κλειδώνεται. αλλά μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Γιατί αυτό σχετίζεται με αυτό που είπαν διάφοροι ομιλητές προηγουμένως για την σύγχυση μεταξύ του αρνητικού και του θετικού καταλόγου και του υβριδικού μοντέλου. Όταν μετακινόμαστε από κατάλογο σε κατάλογο και από μοντέλο σε μοντέλο στις διαπραγματεύσεις, τότε τι γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι αυτό περιπλέκει περιτά τα πράγματα και υποκρύπτονται έτσι κάποια στοιχεία. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι απλό και κατανοητό για όλους όπως ο θετικός κατάλογος που είχαμε στο παρελθόν. Και μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με αυτή την κόκκινη γραμμή για τις δημόσιες υπηρεσίες που ανέφερε η κυρία Ρέντιν και που έχει επαναλάβει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο. Πώς θα μπορούσαμε να πετύχουμε μια πλήρη εξαίρεση των δημοσίων υπηρεσιών. Είπε ο Μάρκους ότι αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι το καλύτερο ως ρήτρα. Μήπως όμως θα έπρεπε να πιέσουμε ώστε να μην πάει αυτό στα παραρτήματα αλλά στο σώμα του κειμένου, στο διατακτικό. Ποια είναι η απόψη σας γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Μαρία. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, παρεμβάσεις. Η παρουσίαση της ε, κυρίας Ρέντινγκ μας παρουσίασε δεξοϊκά τις κόκκινες και τις μπλε γραμμές. Για το μηχανισμό θετικών αρνητικών καταλόγων. Νομίζω είχαμε διάφορε τεχνικές συζητήσεις και επαφέ με την Κομισιόν και είναι αλήθεια ότι οι απαντήσει που λάβαμε είναι ότι το ίδιο είναι είτε αρνητικό είτε θετικό γιατί καταλήγουμε στην ίδια κατάσταση. Αλλά να πω και εγώ, αν είναι το ίδιο, τότε να ακολουθήσουμε την απλούστερη οδό δηλαδή τον θετικό κατάλογο η οποία ως λύση είναι σαφέστερη, πιο περιεκτική και είπαμε στη συζητήση ότι τελικά να καταλήξουμε στην ίδια λύση τότε θα θέλαμε μια πιο διαφανή διαδικασία. Μετά αυτή η ρήτρα αν έχουμε μια κατάσταση όπου εκεί που επιλέξαμε για μια φιλευθεροποίηση κάποιων υπηρεσιών δεν θα μπορούσαμε πρόθεσμα να κάνουμε μια επαναχώρηση σε σχέση με την φιλευθερωποίηση, την απορρίθμιση. Αυτό όμως το επερασπίζουμε με αυτόν τον τρόπο και μου δημιουργεί κάποια προβλήματα γιατί ξέρουμε τι έγινε στο παρελθόν με τις υπηρεσίες και θα πρέπει να διατηρήσουμε τη δυνατότητα επανεξέτασης ορισμών δημόσιας υπηρεσίας που προτείνει μια χώρα όπου γίνεται. Τρίτο ερώτημα. Πώς θα μπορούσαμε στις τωρινές διαπραγματεύσεις να λάβουμε υπόψη μας την ε, προτιμησιακή μεταχείριση που έχει ας πούμε ένα σωτά για τις υπηρεσίε που παρέχει και που τηρεί κάποιες προϋποθέσεις. Παραδείγματος χάρη έχουμε μια υπηρεσία, ε, μια υπηρεσία που παρέχεται από μια επιχείρηση επιχείρηση η οποία τηρεί τις προδιαγραφές για τα εργασιακά οπότε έχουμε τάση να ε, δούμε περισσότερη προτίμηση σε αυτή την επιχείρηση σε σχέση με κάποια άλλη θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, τι γίνεται με τις προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας. Αν τηρούνται αυτές τις προδιαγραφές, τότε θα πρέπει να δίνουμε ε, κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση σε αυτούς που τους τηρούν. Αυτό αφορά την Ευρώπη βεβαίω και το μέλλον τη. Και τέλο, το θέμα τη ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα λεπτό. Στο μέτρο που σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου στην Ευρώπη έχουμε αποδεχτεί ε, την οδηγία που αποδέχεται την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, εργαζομένων, αλλά βλέπουμε και τις δυσκολίες που δημιουργεί. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε ακριβώς ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες που αφορούν την ε, έτσι, λύση σε κάποιες ανησυχίες, επειδή υπάρχει σήμερα ένα social engineering το οποίο εφαρμόζεται και έχουμε καταχρήσεις όσον αφορά το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Μετά, έχουμε και άλλο ένα ζήτημα για τα εργασιακά ακόμα πιο μεγάλο και είναι δύσκολο να το, να το διαχειριστούμε. Θα ήθελα λοιπόν διευκρινήσεις όσον αφορά τη δυνατότητα τήρησης και εφαρμογής του δικαιώματος της εργασίας που έχει να κάνει με τις συλλογικέ συμβάσεις, συλλογικέ συμβάσεις οι οποίες αφορούν συγκεκριμένε επιχειρήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε και αυτό το ζήτημα ώστε σε 10 χρόνια να μην αντιμετωπίσουμε δυσκολίε, οι οποίες δεν θα μα είχαν απασχολήσει και δεν θα είχαμε προβλέψει σήμερα στον αφορά την γενικότητα των εργαζομένων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Χέλμουτ. Έχω ορισμένες ερωτήσεις για τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις των ε, ομιλητών του πρώτου πάνελ. Όπως και η κυρία Αρενά, θέλω πρώτα να ευχαριστήσω την κυρία Ρέντινγκ, η συγγήτρια, για αυτή την ξεκάθαρη αρχική τοποθέτηση. Που όμως με δική στην ερώτηση. Αν μείνουν όλα ε, στο επίπεδο των γκάτς, γιατί χρειαζόμαστε την τίζα. Άρα το ερώτημα είναι, πού ανοίγουμε τους υφιστάμενους κανόνες για τη μελλοντική διαμόρφωση του τομέα του εμπορίου, δηλαδή των υπηρεσιών. Και δεν έχω καταλάβει καλά ως τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως διαπραγματευόμενη, ως μέρος της διαπραγμάτευσης. που περιγράφει τη στάση της. Που μπαίνει σε διαπραγμάτευση με άλλους εταίρους οι οποίοι φέρουν μαζί τους μια διαφορετική κατανόηση για τα θέματα αυτά. Αυτό χρειάζεται διευκρίνηση. Δεύτερη ερώτηση. Είπατε είμαστε ανοιχτοί, inclusive, σε αυτή τη συμφωνία. Άρα, καταρχήν όλες οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και στο μέλλον να την εφαρμόσουν. Πάλι εδώ όμως τίθεται το ερώτημα. Αν έχετε διαφορετική εσωτερική κατανόηση για τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες θα χρειαστεί να γίνει νέα διαπραγμάτευση ή αυτό το συμβατικό κείμενο που θα, στο οποίο θα απορρίξουν οι διαπραγματεύσεις των 24 χωρών θα είναι δεσμευτικό και για τις επόμενες που θα θέλουν να συμμετάσχουν. Τρίτη ερώτηση, και αυτή μου φαίνεται ενδιαφέρουσα. Την έθεσαν και όλοι οι συμμετέχοντες εδώ στο πάνελ, ότι υπάρχουν πολλά τομεακά θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν οριζόντια. Έρχομαι για παράδειγμα στο θέμα της προστασίας των δεδομένων. Πάλι εδώ η διαφορετική ερμηνεία κατανόηση δεδομένων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ενωμένων Πολιτειών που αποτελεί θέμα και στην TTIP. Κατά πόσο λοιπόν μέσα από τις διαπραγματεύσεις στη TISA μπαίνει ένα διαπραγματευτικό θέμα το οποίο θα έχει διαφορετική ρύθμιση στην TTIP ή το αντίθετο. Συζητούμε κάτι στην TTIP όπου πάλι θα υπησέλθει και στην TISA. Πάλι τίθεται εδώ το θέμα της διαφορετικής ερμηνείες, διαφορετική αντίληψη για τα δεδομένα. Και αυτό λοιπόν πρέπει να ξεκαθαριστεί από και διαπαντός για το μέλλον. Τέλος, συμφωνώ με εκείνους που λένε ότι οι κοινοφελείς υπηρεσίες είναι αδιαπραγματεύτε, Απόλυτη κόκκινη γραμμή εκεί. Όμως ως Κομισιόν είπατε ότι προσπαθείτε να βγάλετε απ' έξω το νερό, την παροχή νερού. Αλλά όλα τίθενται επιτάπητος. Όντω τίθενται όλα επιτάπητος. Ή υπάρχει πολύ ξεκάθαρα ένα όριο ότι τα δημόσια αγαθά δεν τα διαπραγματεύεστε. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ο Γιάννικ. Ευχαριστώ του τα μέλη του πάνελ. Εγώ δεν είμαι σκιώδη, ε, εισηγητής για το θέμα της ε, και με ανακουφίζεται γιατί με την TTIP και τη σειτά ήδη οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ε, αντιλαμβάνομαι ακριβώ τη σχέση ανάμεσα στι δύο διαπραγματεύσεις. Ε, δεν αμφισβητώ την αυθεντία της ε, κυρίας Ρέντινγκ. Εγώ όμως δυσκολεύομαι να καταλάβω σε μια διμερή διαπραγμάτευση με την Κορέα, την Ιαπωνία, της ΗΠΑ. Ε, προχωρούμε στις διαπραγματεύσεις και αυτό στη συνέχεια έρχεται στην ΤΙΣΑ ή αντίστροφα. Εγώ δυσκολεύομαι να έχω μια πλήρη εικόνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι διαπραγματεύσεις, αλλά τελικά Έχουμε πάρα πολλές ε, προϊούσες διμερείς διαπραγματεύσεις. Ποια είναι λοιπόν η προστιθέμενη αξία μιας πολυμερούς ε, ε, διαπραγμάτευσης, διότι ουσιαστικά εγώ δεν πιστεύω στην δυνατότητα πολυμεροποίησης, όπως το ονομάζουμε, της συμφωνίας. Άσχετα με αυτά που είπαμε για την Ουρουγουάη, πιστεύω ότι ονειρευόμαστε ότι θα καταλήξουμε σε μια πολυμερή συμφωνία, πολύπλευρη συμφωνία στην με την ΤΙΖΑ, αλλά δεν νομίζω αυτό να υλοποιηθεί. Ε, για ζητήματα εξαιρετικά σημαντικά για τους ε, καταναλωτές ε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε διότι υπάρχει μια ευρύτερη κατανόηση όλων των διακυβευμάτων. Τώρα, θα την ερώτηση και άλλων μελών της Επιτροπής, ε, και απευθύνω την ερώτηση και στα μέλη του πάνελ και στην ε, κυρία Ρέντινγκ. Μιλάμε για την ε, ισχυρή προστασία των δημοσίων υπηρεσιών. Έχουμε μία ρήτρα για την κατοχύρωση και αποκλεισμό των δημοσίων υπηρεσιών. Ποιο δρόμο ακολουθούμε ακριβώς για να προστατεύσουμε τις κοινοφελείς υπηρεσίες. Ε, είχαμε και μια διακοινοβουλευτική συνεδρίαση με τους ομολόγους μας από τον Καναδά προλίγου και ε, μιλούσε ε, κάποιος για την κοινωνική ασφάλιση και μας έλεγε ότι έχει υπάρξει ιδιωτικοποίηση σε διάφορες κομιτείες, σε διάφορες μάλλον περιοχές και του Καναδά και δεν μπορούν να αναιρέσουν αυτό που έκαναν. Ε, η κοινωνική ασφάλιση λοιπόν ε, εντάσσεται στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή στον τομέα της υγείας. Εσείς πώς ακριβώς προσεγγίζετε ένα τέτοιο θέμα. Ε, για σε διαπραγματεύσεις καταλαβαίνω ότι έχει πολλά αποκαλούμενα επιθετικά συμφέροντα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα συνειδητοποιώ ότι θα πρέπει να απελευθερώσουμε και εμείς κάποιες υπηρεσίες ως αντίκρισμα. Μπορεί να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποιους τομείς θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω ανοίγματο σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίσης, όχι μόνο σε εθνικό. Για το Mode 4 ή ένα για ε, τους επιχειρηματίες θα ήθελα να καταλάβω, ε, να μου απαντήσει η κυρία Κλάρκ, αν θεωρεί ότι ελοχεύει κινδύνους και το Mode 1 για τον ανταγωνισμό προς τα κοινωνικά πρότυπα κατά την διασυνοριακή ανταλλαγή υπηρεσιών. Πρόεδρος, και εγώ μια ερώτηση, ιδίως για τον κύριο Καγιεύσκη. Το ζήτημα της ε, συνέπειας. Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει αυτή η συνοχή μεταξύ της ΤΙΖΑ και για παράδειγμα της ΣΕΤΑ. Παραρτήματα 1 και 2 που προβλέπουν ειδικέ εξαιρέσεις για επιμέρους χώρες μέλη. Υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα σε αυτές. Και ποια θα είναι η επιρροή της ΤΙΖΑ σε αυτές τις διμερείς σχέσεις, διμερείς συμφωνίες καλύτερα. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο για τρία λεπτά σου σε καθέναν από τους ε, εμπειρογνώμονες και θα αρχίζουμε με την ίδια σειρά, πρώτα δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις των μελών για τη διαφάνεια. Κάναμε πάντο το δυνατό και στην ιστοσελίδα μας τα δημοσιεύουμε όλα. Δεν μπορούμε να ανακάσουμε τις χώρες μέλη να κάνουν το ίδιο. Το ίδιο ήταν και στις ε, συμφωνίες, του ΠΟΕ. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νορβηγία και Ελβετία έχουν ε, ε, δημοσιεύσει τις προσφορές τους στην ΤΙΣΑ. Τώρα, αρνητικός και θετικός κατάλογος. Η υβριδική προσέγγιση βασίζεται σε μια θεσμική συμφωνία από την αρχή. Υπήρχαν και εκείνοι, όπως εμείς, που έλεγαμε ότι θέλουμε την αρχιτεκτονική GATS, δηλαδή θετικό κατάλογο. Για άλλους αρνητική, αρνητικός κατάλογος ήταν μέρος του κεκτημένου για ορισμένε χώρες. Αυτό φαίνεται την πιο κοντά στον ΚΑΤ. Έχουμε πρόβλημα, ρωτήσατε, με τα εργασιακά δικαιώματα, με την κινητικότητα των εργαζόμενων όχι για προσωρινή κινητικότητα. Έχουμε ωστόσο επιφύλαξη στην προσέγγιση μας, στην προσφορά μας μάλλον, θα τη βρείτε και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιφύλαξη που λέει ότι στην περίπτωση προσώπων που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκατασταθούν, ισχύουν οι διάφορες ρυθμίσεις, θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις, για παράδειγμα, για διάρκεια παραμονής για ελάχιστους μισθούς, αμοιβέ κλπ. Έχουμε λοιπόν μια ξεκάθαρη επιφύλαξη που λέει ότι σε ό,τι αφορά ελάχιστους μισθούς και ελάχιστες υποχρώσεις που απορρέουν από συλλογικές συμβάσεις κτλ. Αυτά ισχύουν. Αυτά μπαίνουν και σε όλες τις συμφωνίες για το εμπόριο υπηρεσιών. Πάμε πέρα από τον ΚΑΤΣ. ρωτήσατε και ποια είναι η σχέση plurilateral-multilateral που μεταφράζεται ελληνικά πολυμερής και στα δυο. Αν έχουμε κάποια στιγμή μια κρίσιμη μάζα θα την φέρουμε, θα φέρουμε στο πλαίσιο του ΠΟΕ και τότε θα ισχύει και για χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν σήμερα. Μπορούμε να φέρουμε τώρα υπηρεσίες που σε κάποιες χώρες είναι ιδιωτικές στο πλαίσιο των δημοσίων κοινοφιλών υπηρεσιών. Ναι, Νομίζω μπορούμε να μονοπολίσουμε μια υπηρεσία που σήμερα είναι ιδιωτικοποιημένη, μπορούμε να την φέρουμε σε κρατικό μονοπόλιο στην βάση των υποχρεώσεων που έχουμε ήδη αναλάβει. Και προσπαθήσαμε να το εξηγήσουμε τεχνικά αυτό και σε άλλα πλαίσια. Νομίζω ότι έληξαν τα τρία μου λεπτά. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ. Εσείς κύριε καθηγητά τώρα. Η διαφάνεια είναι σημαντική πράγματι. Το γεγονός ότι οι προσφορές είναι διαφανείς, αυτό δεν είναι ίσως τόσο σημαντικό γιατί οι προσφορές βασίζονται σε συμφωνίες που έχουν γίνει από πριν. Αυτό είναι γνωστό. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τα αιτήματα, τα requests. Γιατί δεν βλέπουμε και αιτήματα της Ένωσης που και αυτή ζητεί πράγματα. Επίσης κεφάλαια, ρυθμιστικά κεφάλαια. Ακούω τον κύριο Μπανές που λέει ότι η Κομισιόν του τα έχει διαβιβάσει. Σε αυτόν και εγώ έχω δει ορισμένα βέβαια υπό συνθήκε αυστηρής εμπιστευτικότητας. Αλλά διαρωτώ με, αν δείτε την πρόταση για την Τουρκία, δεν είναι τίποτε ε, μυστικό κρατικής ασφάλειας. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν. Είναι περίπλοκα θέματα. αν είναι δηλαδή ε, ζητήματα ε, ρύθμισης των ασφαλιστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας κλπ. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν ε, καθίστανται δημόσια ως κανόνα και όχι βεβαίως ως παραχώρηση κάποιας χάρης ιδιαίτερης. Τώρα, για την επαναδιαπραγμάτευση. Το σχέδιο πρότασης που είδα δεν περιλαμβάνει τις σχετικές ρυθμίσεις GATS, αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσει να υπαχθεί και αυτό. Το χρονόμετρο βλέπω δεν λειτουργεί, δηλαδή μπορώ να μιλώ όσο θέλω. Συνεχίζει. Για το θέμα της συνοχής. Εδώ είναι δύσκολο το πράγμα. Βέβαια μπορεί κανείς να αντιγράψει διατάξεις του ΓΚΑΤΣ και να πει ότι είναι το ίδιο. Το ζήτημα είναι πόσο συνεκτικές είναι αυτές οι δεσμεύσεις. Είναι πολύ τεχνικό το θέμα αυτό. Μόνο όταν δούμε τις σχετικές δεσμεύσεις θα μπορέσουμε να κρίνουμε. Ακόμα δεν έχω πλήρως μελετήσει τις δεσμεύσεις της ΕΤΑ. Μπορούμε να μονοπολίσουμε πώς προστατεύουμε τις κοινοφελείς υπηρεσίες. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Και μου φαίνεται ακόμη ότι για να προχωρήσουμε χρειάζεται όχι μια συνολική ρήτρα, μια catch-all phrase η οποία θα λέει ότι τα βάζει όλα μέσα. Τα βήματα που έχουν γίνει στη ΣΕΤΑ είναι σημαντικά, αλλά πρέπει να συνεχιστούν τα μέτρα αυτά. Η ΠΕΝ είπε ήδη ότι και ο ορισμός των δημόσια χρηματοδοτούμενων μπορεί να μην αρκεί. Μπορούμε να τις επαναφέρουμε στο μονοπόλιο, ναι. Ε, εάν ο τομέας καλύπτεται από την εξαίρεση για τις δημόσιες κοινοφελείς υπηρεσίες, ναι. Αλλά πάλι αυτό είναι ανοιχτό σε συζήτηση. Και αυτή είναι η τελευταία μου φράση. Στη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη υπάρχει, ε, περιλαμβάνεται μια ενδιαφέρουσα τεχνική. Υπάρχει θετικός κατάλογος και για κάθε τομέα που θα πρέπει να ισχύει η προστασία των κοινοφιλών υπηρεσιών μπαίνει και μια υποσημείωση. Είναι χρήσιμη προσέγγιση αυτή. Δεν ξέρω βεβαίω αν υπάρχει κανένα λάθο, ε, αλλά ο τομέα τη παιδεία δεν έχει υποσημείωση. Άρα προφανώ δεν εντάσσεται στι δημόσιε κοινοφιλές υπηρεσίε. Σας ευχαριστούμε κυρία yeah, I would say certainly it's... Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Σημαντικό είναι να υπάρχει αυτή η γνώση. Τα μικρά, τα μεγάλα στοιχεία, υποσημειώσεις, όπως είπε και ο Μάρκ, να μην έχουμε κάτι το οποίο ισχύει για τα πάντα. Είδα το κείμενο και τις γενικές εξαιρέσεις. Νομίζω ότι δεν είναι αδυνατόν να επεκταθούν. Να μην πούμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για θέσπιση μια ηθικής ας πούμε παραπομπής. Είπε και ο Ιγνάθιο κάτι προηγουμένως για, τις, για τους κανονισμούς. Όμως αυτούς τους κανονισμούς χρειαζόμαστε για τις δημόσιες υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό Πρέπει λοιπόν να γίνουν και άλλες συζητήσεις. Να αναφερθώ σε κάποια θέματα που ανέφερε συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλια που σημείωσα και θα έρθω σε επαφή μαζί σας για να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες γιατί τώρα δεν έχουμε χρόνο αλλά για την εξαίρεση των δημοσίων υπηρεσιών βεβαίως όμως οριζοντίως το κείμενο αφορά όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και θα ήθελα να περιλάβουμε εδώ στι δημόσιες και τι κοινοφιλεί υπηρεσίε. και να δούμε και το κεφάλαιο για του δημόσιου διαγωνισμού, ε, όπω είπε και η κυρία Ρένα έχουμε τι συμβάσει του Παγκοσμίου Οργανισμού Εργασία. Στι ρυθμίσει μα υπάρχει όντω παραπομπή στον Παγκοσμίο Οργανισμό εργασία και υπάρχει και μια ρήτρα η οποία ελπίζω θα περιληφθεί σε όλες τους δημόσιους διαγωνισμούς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις συλλογικέ δηλαδή συμβάσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχουν θέματα που αφορούν την εργασία στην Ευρώπη. Το δικαστήριο έχει επιληφθεί κάποιων αυτών των θεμάτων. Αφορά τα συνδικάτα και νομίζω ότι οι καλοί εργοδότες ε, θέλουν να προστατεύουν τους εργαζόμενους τους, να τους ε, πληρώνουν σωστά ώστε ώστε, αυτό, ώστε αυτοί να αποδίδουν. Και αυτό πρέπει να είναι θέμα συνένεση μεταξύ μα. Έχουμε και τα περιβαλλοντικά κριτήρια που έχουμε σημαντική αναγνώριση του γεγονότος ότι μπορούμε να, μην χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία των δημοσίων ε, διαγωνισμών. Έχουμε τη διακριτική ευχέρεια στο άρθρο 4 που αναγνωρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση για τη ΟΤΑ. Ένα τελευταίο στοιχείο η σχέση μεταξύ των διαφόρων συμφωνιών. Νομίζω ότι δεν το συζητήσαμε αρκετά τώρα, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε μελλοντικά. Νομίζω υπάρχουν πάρα πολλές διαπραγματεύσεις επιμέρους και θα έχουμε νομίζω στενές επαφές για το μέλλον της εμπορικής πολιτικής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούσαμε και κάποια σχόλια για το θετικό και το αρνητικό κατάλογο είπε το Κοινοβούλιο ότι δεν μπορεί να αποτελεί προαπαιτούμενο αρνητικό κατάλογο ε, για τον επόμενο γύρο. Εμεί τι κάνουμε όμω με τι άλλε χώρε στο εμπόριο σε σχέση με του αρνητικού ε, καταλόγους, τι θέλουμε να κάνουμε ακριβώ με τι γειτονικέ μα χώρε, Πολλά πρέπει να πούμε εδώ. Εγώ σημείωσα όλα αυτά τα θέματα πάντω και προσβλέπω σε περαιτέρω συζήτηση μαζί σα γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Βεβαίως είμαστε υπέρ μεγαλύτερης διαφάνειας. Η εντολή που θα έχουμε σύντομα τονίζει ακριβώς το δημόσιο χαρακτήρα και υπάρχει και ανταπόκριση από τις ΕΠΑ που το διατυπώνουν πιο ήπια. Νομίζω ότι Όλοι θέλουμε να αποφύγουμε χρονοβόρες ε, διαδικασίες και θέλουμε βέβαια όλοι οι χώρες να δημοσιεύουν τις προσφορές τους, τις αντιπροτάσεις τους και θα πιέσουμε γι' αυτό. Για το θετικό και αρνητικό κατάλογο τώρα. Ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να υπάρχει αρνητική λίστα είναι για μια επιχείρηση. Ας πούμε, αν δούμε τις αντιπροσφορές της ΣΥΤΑ. Ξέρετε ότι ό,τι περιλαμβάνεται, από αυτά περιλαμβάνονται, τι είναι εφικτό και τι όχι. Αν δούμε ένα το θετικό κατάλογο, όπου μια χώρα δεν περιλαμβάνεται δεν είναι ότι αποκλείεται, είναι ότι σημαίνει ότι δεν έχει αναλάβει ε, δεσμεύσει και ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά να δούμε τι μπορεί να γίνει. Για το πώς θα προχωρήσουμε τώρα, για την κινητικότητα. Μιλάμε για προσωρινή κινητικότητα. Το Διεθνές Εμπόριο Υπηρεσιών αφορά συνήθως τη σχέση μεταξύ δύο επιχειρήσεων. Χρειάζεται η επιχείρηση να επισκεφθεί ας πούμε τις ιατρικές της, να έχει επαφή με τους πελάτες της κτλ. Δεν έχει σχέση με την μη τήρηση ε, των ε, προβλεπωμένων για τις συλλογικές συμβάσεις ας πούμε. Νομίζω ότι όλες οι υποσημείες του κείμενου είναι σαφείς επ' αυτού και θεωρούμε ότι στο τίστα δεν θα έχουμε διαφορές επ' αυτού. Για τις μόσιες υπηρεσίες δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο φόβο. Θέλουμε η ΤΙΣΑ να επικεντρωθεί στο διεθνέ εμπόριο, στις, στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών. Και σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε τι διεθνεί εμπορικέ υπηρεσίε, υπάρχει και αντίστοιχη επιτροπή. Έχουμε 150 δις πλεόνασμα ε, όσον αφορά τις εμπορικές υπηρεσίες, δηλαδή ε, τρει τελικά. Γι' αυτό μιλάμε. Αυτό πρέπει να αυξηθεί. Δηλαδή αυτή η επιτροπή δεν αφορά τι δημόσιε υπηρεσίε, αλλά τι ιδιωτικέ υπηρεσίε. Αν θέλετε καλύτερη διατύπωση εντάξει, αλλά α το συζητήσουμε και να επικεντρωθούμε στο εμπόριο. Για τη διατύπωση που είπε ο Μάρκου το τι αναφέρεται στο, ΣΥΚΑ, στο ΣΥΤΑ είναι αρκετά καλό και γενικόλογο ω διατύπωση και καλύπτει νομίζω και διασκεδάζει τι ανησυχίε που υπάρχουν για τι δημόσιε υπηρεσίε. Τώρα για την προστόμενη αξία τη ΤΙΣΑ και την ε, σύγκριση με τις άλλες πολυμερίες Η πολιτική, συγγνώμη, η προσθέμενη αξία ακριβώς είναι αυτό το θέμα της προστασίας, της περισσότερης προστασίας που θα προσφέρουν περισσότερες χώρες. Βεβαίως πρέπει να προχωρήσουν παραπέρα οι πολυμερίες και η ΤΙΖΑ αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο ώστε να έχουμε βεβαιότητα και ασφάλεια ε, διεθνώς σε αυτό. Ευχαριστώ. και στην Επιτροπή μας οφείλουμε να φροντίζουμε για τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και είμαστε εκπροσωποί τους εν τέλει. Ας έλθουμε τώρα στο δεύτερο πάνελ για επιμέρους τομείς που συζητήσα πρώτα για τις τηλεπικοινωνίες με τον κύριο Λάρι Στόουν της Βρετανικής Τελεκόμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα. Υποστηρίζει η British Telecom μια αμοιβαία προσέγγιση, win-win, αμοιβαίως επικερδούς για την ΤΙΣΑ ε, στα πλαίσια των πολυμερών διαπραγματεύσεων που έχουν ολοκληρωθεί, ε, των διμερών διαπραγματεύσεων ε, μάλλον με την Κορέα ή την Ιαπωνία ή των πολυμερών με την Μέρκοσουρ. Είναι περίπλοκο το ζήτημα, θα επανέλθω σε αυτές. Βασικός φορέας είναι η BT, δραστηριοποιούμαστε σε 170 χώρες στον κόσμο ε, και ε, έχουμε, προσφέρουμε υπηρεσίες πληροφορική σε πολυεθνικές, σε κυβερνήσεις, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ε, προσφέρουμε άμεσα υπηρεσίες ή μέσω ενδιαμέσων και μερών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις της ΤΙΣΑ. Έχουμε μια βασική ραχοκοκαλιέβαση, το βασικό μας δίκτυο δίκτυο καλύπτει σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου. Ε, για ποιο λόγο υποστηρίζουμε τις διαπραγματεύσεις της ΕΠΕ. Πρώτον, πιστεύουμε ότι είναι βασική δύναμη ε, στις υπηρεσίες ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μου και νομίζουμε ότι αυτό δημιουργεί ένα ικανοποιητικό δυναμικό ανάπτυξης ε, και μπορούμε να εξάγουμε το νόμισμά μας και να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα ηλεκτρονικού εμπορίου και να εξαγάγουμε το μοντέλο μας. Επίσης, είπαμε ότι το 70% του παγκοσμίου παγκοσμίου εμπορίου στις υπηρεσίες προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι νομίζουμε ότι θα βοηθηθεί η οικονομική ανάκαμψη με την διεύρυνση, την εξαγωγή του μοντέλου μας προς τρίτες χώρες. Στη συνέχεια ε, πιστεύουμε ότι σε σχέση με τις χώρες του ΑΣΕΑΝ στην Ασία μπορούμε να ενισχύσουμε την, υπηρεσία, την παρουσία μας ε, στην Ασία. Στη συνέχεια ε, θεωρούμε ότι μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη η ροή πληροφοριών και υποδομή των τηλεπικοινωνιών με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Τέσσερα, ε, μπορούμε να έχουμε μια ευθυγραμμισμένη πρόσβαση στην αγορά και τυποποιημένους όρους ε, ε, πρόσβασης ε, για τους ε, πελάτες των επιχειρήσεων και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Πέμπτον, ελπίζουμε ότι η ΤΙΣΑ μπορεί να ενισχύσει την ανοιχτή και απρόσκοπτη διασυνοριακή ροή πληροφοριών, ενώ ταυτόχρονα θα συμφωνήσω, όπως είπε και η κυρία Ρέντινγκ, τα τοπικά τα καθεστώτα προστασίας ε, των δεδομένων με βάση και των ε, αυτών που έχουν κατοχυρωθεί στην ε, Συμφωνία GATS. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, πιστεύουμε ότι χάρη στην ΤΙΣΑ μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικότερα πιο ανοιχτά καθεστώτα για την, τις δημόσιες προμήθειες, κυρίως στον τομέα της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών. Μπορούμε να κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες τους φραγμούς, μειωμένη πρόσβαση, ε, περιορισμένη πρόσβαση με τα ανώτατα όρια ε, και τρίτον ε, και τοπικές ρυθμίσεις λόγω εθνικών νομοθεσιών κατά των τραστ. Όσοι μετέχουν στις διαπραγματεύσεις της συνειδητοποιούν ότι δημιουργούν προκύπτουν διαρκώς αλλαγές ε, ε, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια ανεξάρτητη νομοθεσία παραδείγματος χάρη για τη προστασία των δεδομένων κάτι που θα ήταν και υποφελής για το διεθνές εμπόριο. Αποτελεσματική νομοθεσία έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για την διασυνοριακή αλλά και για την εγχώρια παροχή υπηρεσιών. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να εμβαθεί την ψηφιακή της αγορά και υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να έχουν την ίδια ποιότητα τα υπηρεσιών στις συνδέσεις που έχουν ε, σε διάφορες χώρες και προτιμούν να έχουν έναν παρόχο για το υπολογιστικό νέφος ε, ή για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ε, ή στον τομέα του συνεργατικού σχεδιασμού παραδείγματος χάρη. Θέλουν λοιπόν επίσης να αναβαθμίσουν την διαδικτύωση στο εσωτερικό μιας πολυεθνικής εταιρείας και να προωθήσουν την καινοτομία, την έρευνα και την καινοτομία σε τομείς, όπως σας είπα, του, ε, της ε, συνεργατικής επιχειρηματικότητας ε, και την μετάβαση στο διαδίκτυο 4.0 βελτίωση της διασυνδεσιμότητας ε, λοιπόν βλέπουμε πως ε, η ισότιμη πρόσβαση σε βασικές υποδομές, ε, κατοχύρωση της διαφάνειας και πλήρη εικόνα των νομοθετικών ρυθμίσεων είναι κάτι που επιθυμούμε η ΕΠΑ, η Ιαπωνία, η Νορβηγία και άλλες χώρες της όπως η Χιλή έχουν ξεχωριστή νομοθεσία για την, ένα θεμελιώδη λίθο της πρόσβασης στην ισότιμη παροχή υπηρεσιών. Στη είπανε για να πάρουμε ένα παράδειγμα γιατί έχουν υποδειγματικό ρόλο. Ε, θα ήθελαν ε, να επέμβουν σε αυτό το τομέα και ε, αυτό θα αγγίξει και άλλες ε, χωρίς που ενδεχομένω ε, στη συνέχεια να ε, προσχωρήσουν σε σχέση με τα βασικά τηλεπικοινωνιακά πρότυπα στα μέσα του 19... που εγκρίθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Φυσικά μετά την Τόχα υπάρχουν πάρα πολλοί, πολλοί διάλογοι που και ειδικότεροι βλέπουμε πως η αξία ε, θα είναι περίπου 90 δις ε, ε, δολάρια ε, και συνειδητοποιούμε πως ε, το ενδεχόμενο όφελος για τη ΣΥΠΑ θα ήταν 160 δις σε σχέση με τις επενδύσεις και φυσικά όλα αυτά σημαίνουν και νέες θέσεις εργασίας. Ένα κάτι τελευταίο να προσθέσω, Πρόεδρε, φυσικά ε, έχουν αποτύχει οι διάφοροι γύροι της Ντόχα στα πλαίσια του ΠΟΕ. Έχουμε άλλους πολυμερείς διαλόγους ε, και βλέπουμε ότι ένα βασικό πρόσκομα είναι ε, η διευθέτηση των διαφορών ε, ανάμεσα στους επενδυτές και στα κράτη. Είναι, λένε και μεγαλύτερη πρόκληση αυτό και θα είναι σημαντικός ο ρόλος της ΤΙΖΑ αυτό. Ποιος θα είναι ο ρόλος του ΠΟΕ, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημείο εκαθάρισης ε, σε ένα οριζόντιο επίπεδο για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στο Δουβλίνο. Πριν από ένα χρόνο μίλησα για αυτά τα εμπορικά ζητήματα και οι, οι ε, ε, φάνηκε να υιοθετούν μια τέτοια ιδέα. Δεν ξέρω αν θα, μπορούσε, θα μπορούσαμε να προωθήσουμε μια τέτοια πρόταση, αλλά θα μπορούσαμε τουλάχιστον να την εξετάσουμε. Ευχαριστώ πολύ για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών λοιπόν. Ας έρθουμε τώρα στις ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Edward Bowles, Public Affairs Europe, από μια τράπεζα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τις και τους συναδέλφους σας για την ε, γραμματεία σας που μας διευκόλυνε να περάσουμε. Εμείς είμαστε, έχουμε την έδρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 90% της ε, business μας γίνεται με χώρες ε, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Έχουμε λοιπόν πραγματικά εμπόδια που αντιμετωπίζουμε. Τούτου λεχθέντος είμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις αγορές αυτές. Θα επανέλθω λοιπόν σε ορισμένες συγκεκριμένε παρατηρήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες χρηματοπιστωτικών χαρακτήρα. Υποστηρίζουμε την ΤΙΣΑ, ναι, υποστηρίζουμε ορισμένες, με ορισμένες επιφυλάξεις. Θα επανέλθω. επανέρχομαι στην αρχική τοποθέτηση της κυρίας Ρέντινγκ που ήταν απόλυτα σαφής. Θα κάνω τρία πρώτα σχόλια για την διαφάνεια πρώτα και το αίτημα να μην λάβει το χαρακτήρα της TTIP ή TISA. Έχω και άλλες ιδιότητες, είμαι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την TTIP ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η TTIP έχει κάνει μεγάλη ζημιά, τεράστια ζημιά, τεράστια ζημιά λόγω του ότι δεν υπήρξε διαφανής εξ αρχής. Αν δείτε την εντολή 19 σελίδων για την TTIP, δεν προβλέπει απολύτως τίποτα την αδιαφάνεια αυτή επί 1,5 χρόνο. Έτσι λοιπόν είμαι απόλυτα υπέρ της ε, αποφασιστικότητας της κυρίας Μάλμστρομ να καταστήσει διαφανή την ε, δημόσια την ε, διαπραγματευτική εντολή. Και το ίδιο και για την ΤΙΣΑ. Μα δεν είναι απόρριτα πράγματα αυτά, δεν είναι απόρριτες διαπραγματεύσεις και δεν πρέπει έτσι να αντιμετωπίζονται. Τίποτα από αυτά δεν μπαίνει σε κάποιο ε, χώρο απορρίτου. Το ίδιο σε ό,τι αφορά έγγραφα θέσεων. Η Κομισιόν έχει εκδώσει τον Ιούλιο του 2013 ένα έγγραφο που περιλάμβανε τα παρατήματα του Γκάτς και το Μνημόνιο Συμφωνίας και μετά αυτό επεκτάθηκε και ελπίζω ότι η Wikileaks και μάλιστα χαίρομαι που η Wikileaks δημοσίευσε τα υπόλοιπα που συζητήθηκαν και στον 11ο γύρο πριν από 10 ημέρες στη Γενέβη. Έχει γίνει λοιπόν πρόοδο σχετικά. Πάλι όμως, όταν δείτε το σχέδιο της Wikileaks, δεν βλέπετε ούτε σε αυτό το σχέδιο τίποτε που να μπορεί να αρθεί σε ύψος ε, εθνικής ασφάλειας έτσι ώστε ε, να δικαιολογεί την έλλειψη διαφάνειας. Έτσι λοιπόν για το πρώτο πράγμα που είπατε έχετε απόλυτο δίκιο όσο μεγαλύτερη διαφάνεια τόσο το καλύτερο και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην αρχίσουμε και τώρα έστω και με καθυστέρηση να τα κάνουμε διαφανή. Δεύτερο τώρα για να γίνει η τίσα πολυμερής. Ε, αυτό πρέπει να είναι πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προ 18 μήνου οι Ενωμένε Πολιτείε που ανθίσταντο στην, στον δεχόμενο να μπει η ΔΟΚ μέσα σε ένα πολυμερές πλαίσιο. Η Κομισιόν ωστόσο έστησε τα πόδια, ήταν αποφασισμένη, είπε ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει στην ΤΙΣΑ θα πρέπει να μπει σε ένα πλαίσιο πολυμερές. Multilateralized. Λοιπόν, αυτό συμφωνήθηκε τελικά. Έχουμε λοιπόν κάτι το οποίο θα είναι δυνατόν να μπει σε ένα πλαίσιο πολυμερές στο μέλλον. Τώρα, πού βρισκόμαστε και έρχομαι εδώ ε, στην υποστήριξή μου για την Τίσα. Η Τίσα στον πυρήνα της είναι, έχει ως στόχο να κάνει δεσμευτική τις, δεσμευτικές τις τρέχουσες πρακτικές και το μηχανισμό standstill που έχετε όχι μόνο στο σχέδιο για τις χρηματοδοτικές υπηρεσίες αλλά και σε άλλα σχετικά έγγραφα. Ακόμα όμως και ο μηχανισμός standstill δεν θα καθοριστεί, δεν θα οριστεί μονάχα από μη συμμορφούμενες πρακτικές. Ορισμένα μέρη των διαπραγματεύσεων θα προβάλλουν επιφυλάξεις που θα τους επιτρέπουν να υπαναχωρήσουν από τις υφιστάμενες ήδη πρακτικές. Ακόμα και ο μηχανισμός standstill, δηλαδή στην καρδιά του, δεν, ήταν, δεν απεδείχθη να είναι αυτό που είχαν ελπίσει από την αρχή των διαπραγματεύσεων. Διότι το νόημα της ΤΙΣΑ είναι να πούν ότι ο αριθμός χωρών που θέλουν να προχωρήσουν πέραν των δεσμεύσεων που έχουν λάβει από τον ΚΑΤΣ και άλλες που δεν τα έχουν δεχτεί ακόμα αυτά, ήδη υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις ΚΑΤΣ. Ας τα βάλουμε λοιπόν σε ένα ενιαίο κείμενο συμφωνίας για να έχουμε ένα κατόφλι. Όμως στις χρηματοπιστευτικές υπηρεσίες γνωρίζουμε ότι ένας αριθμός από τους συμμετέχοντες θέλουν να προβάλλουν επιφυλάξεις, να τις καταθέσουν δηλαδή. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα διαπραγματευόμενα μέρη τηρούν ρωμαλαία θέση και ζητούν απόλυτη εξειδίκευση απέναντι σε αυτά τα πιο διστακτικά διαπραγματευόμενα μέρη. Αλλά δεν είναι ισότιμος ο αγώνας. Τώρα, ειδικότερα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οροφές στην δυνατότητα να κατέχουν οι επιχειρήσεις ε, μετοχές των θηγατρικών τους στην Αλλοδαπή είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα σχετικό ερωτηματικό και ο στόχος πρέπει να είναι να καταργηθούν και πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο των ετοιμάτων μας. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα της ενισχυμένης subsidiarization, γιατί ορισμένες από τις χώρες, μέλης, χώρες ε, αυτές εμποδίζουν ορισμένες χώρες να συναλλάσσονται με τις ομολογίες τους. Γι' αυτό εταιρείε χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μπορούν να λειτουργήσουν μόνο εφόσον έχουν μια θηγατρική επιτόπου που σε ορισμένε περιπτώσεις είναι στην περίπτωσή μας για παράδειγμα εδώ και 150 χρόνια στην ε, Ινδία ή 150 χρόνια στην Κίνα ή στην Ταϊβάν. Υπάρχει όμως μια τάση προς ενίσχυση αυτής της θηγατρικότητας που ωστόσο θα έχει αντιπαραγωγικό αποτέλεσμα όσον αφορά την αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και διαμεθοριακά, που είναι τόσο σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παλαιότερα, εσείς κύριε Ρέντινγκ, είχατε ταχθεί υπέρ της ε, προστασίας των δεδομένων. Στα σχέδια των εγγράφων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δεν βλέπω να υπάρχει τίποτε που να υπονομεύει τους στόχους που είχατε θέσει τότε αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι τα, μέσα, τα μέτρα μέσα των οποίων προσπαθούν να χειραγωγήσουν την αγορά και την προστασία δεδομένων σε ορισμένε περιπτώσει. Αυτό που είδαμε και στην Free Trade Agreement με την ε, Κορέα είπε στην Κορέα αντιλαμβανόμαστε την, το ιστορικό με ό,τι φαίνεται οι, ε, οι Ιάπωνες παρέβησαν κανόνες στο παρελθόν, αλλά αυτό είναι παρελθόν. Τώρα πρέπει να επιμείνουμε ότι θα λειτουργούν σωστά οι άξονες διακίνησης των δεδομένων, data hubbing δηλαδή. Οι δικοί μας, οι δικοί ρυθμιστές μας απαιτούν να έχουμε και backup systems. Αν έχετε ένα σύστημα onshore θα πρέπει να το έχετε και offshore για να μπορείτε να υποστηρίξετε ένα σύστημα που ενδεχόμενα θα πέσει και υπάρχουν ε, οικονομικοί λόγοι για να υπάρχει και το data hubbing. Κύριε Πρόεδρε, πριν να ολοκληρώσω μια τελευταία λέξη, βέβαια δεν έχει σχέση απαραίτητα με την TTIP. Σας συγχαίρω όμως για το σχέδιο εκθέσεώ σα που συζητείτε σήμερα το απόγευμα και ιδίως για την πρώτη παραγραφή που έχει σχέση με τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε και που συνδέεται την υπηρεσία των προσβάσεων σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ και την συνεργασία. Για τους λόγους που αναφέρετε στην παραγραφό σα, που λέτε ότι αν υπάρχει υπάρχουν μάλλον μη συνεκτικά ε, νομοθετικά πλαίσια ανοίγεται το χώρο για το arbitrage και επομένως για την οικονομική αστάθεια. Είναι σημαντικό λοιπόν όλοι μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθειά της να φέρει τις ΗΠΑ γύρω από, το, από την Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Να υπάρχει δηλαδή εντολή για να μειωθεί το ε, εύρος του αρμπιτράζ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. τελευταίο τομέα οι ταχυδρομικέ υπηρεσίες, ο κ. Σαδωράκης, υπεύθυνο Πολιτική και επιμελητία από την Uni Global Union Europe. Παρακαλώ. Καλημέρα κυρίε και κύριοι. Εξέχοντα μέλη του Κοινοβουλίου. Εκπροσωπώ τον τομέα επιμελητία και ταχυδρομικών υπηρεσιών της Uniglobal Union Europe με πολλές επιχειρήσεις και εργαζόμενους παγκοσμίω. Όπως επίσης και τα κούριες και άλλες επιχειρήσεις επιμελητίας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω στο Κοινοβούλιο σήμερα για αυτό το σημαντικό ζήτημα για τα μέλη μας που προκαλεί ανησυχίες. Όπως και οι συνάδελφοι και από άλλες οργανώσεις, εμείς στείλαμε διάφορες επιστολές ζητώντας την αποχώρηση από τις ε, συζητήσεις και την καταγγελία. Η απάντηση μου λοιπόν στο ερώτημα είμαστε υπέρ της είναι αρνητική. Όχι. Επαναλαμβάνουμε τις επιφυλάξεις μας στις ε, διαπραγματεύσεις για την διάβρωση των δημοκρατικών διαδικασιών και για τη μυστικότητα των διαπραγματεύσεων και νομίζω αυτό που άκουσαν σήμερα το επιβεβαιώνουν. Μιλώντας εξ ονόματο των μελών μας στον τομέα των υπηρεσιών επιμελητίας και τεχνικών υπηρεσιών έχουμε εμπειρία ε, δύο δεκαετιών φιλελευθερωποίηση στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και είδαμε τα αποτελέσματά της που είναι απτά και αρνητικά. Η φιλελευθερωποίηση στον τομέα αυτό είχε ολέθριες επιπτώσεις ε, στην Λατινική Αμερική, στην Ασία και ξεκινά να έχει τις ίδιες επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για γενιές οι ταχυδρομικές υπηρεσίες βρισκόταν στο επίκεντρο οικονομικών συστημάτων χωρών. Παρήχαν υποδομή και δίκτυα επιτρέποντας ε, στους πολίτες να επικοινωνήσουν και στις επιχειρήσεις να προοδεύσουν. Σήμερα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των οικονομιών μας και των κοινωνιών μας. Αποτελούν ένα κύριο ε, δίκτυο επικοινωνίας βασιζόμενο σε αυτή την ε, αρχή της κοινοφελούς υπηρεσίας και θα επανέλθω αυτό στη συνέχεια της ομιλίας μου. Ως ε, οργάνωση θεωρούμε ότι η πρόσβαση σε ε, αυτές τις, σε υπηρεσίες πρέπει να ασφαλίζεται από την δημόσια διακυβέρνηση. Και τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης, φιλελευθερωποίηση όμως η οποία έχει διαταράξει τις οικονομίες όσον αφορά την παροχή αυτών των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Δυσκόλεψε τους εμπλεκόμενους φορείς στην παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών ώστε αυτές να παρεχόνται με οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο. Η ιστορία λοιπόν της φιλελευθερωποίησης αυτών των υπηρεσιών αποτελεί στην ουσία διάβρωση της υποχρέωσης για υπηρεσίες παροχή υπηρεσιών καθολικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπόσχεται καλύτερες ταχυδρομικές υπηρεσίες με χαμηλότερες τιμές και δυστυχώς πρέπει να προσθέσω ότι αυτό δεν έχει υλοποιηθεί. Αντίθετα, βλέπουμε να υπάρχει, βλέπουμε να υπάρχει κατακαιρματισμός της αγοράς και να εξαιρούνται διαφοροί από τις υποχρεώσεις ενώ ταυτόχρονα αποφελούνται στο ακέραιο από τις οικονομικές ευκαιρίες. Επίσης, έχει δοθεί βοήθεια στα διάφορα μονοπόλια μέσω διαφόρων επιδοτήσεων. Ο ανταγωνισμός σήμερα αφορά κυρίως το πεδίο των τιμών που παραμένουν ε, πολύ, πολύ χαμηλές όσο και οι μισθοί και απολαβές των εργαζομένων. Και βεβαίως αυτό αφορά και τους καταναλωτές γιατί δεν έχουμε καταφέρει να ανταποκριθεί στην υποχρέωση για χαμηλέ τιμές και υψηλή ποιότητα. Επίσης, η φιλελευθερωποίηση ήταν καταστροφική για τους αποσχολημένους στον τομέα. Σημαίνει ότι είχαμε απώλεια θέσεων εργασία στον τομέα και κυρίως επιδίνωσε τι συνθήκες εργασίας στον τομέα της επιμελητίας, ταχυδρομικής επιμελητίας, το, το πλεονέκτημα αφορά συνήθως την περικοπή στις τιμές αυτό βέβαια οδήγησε όλους τους εμπλεκόμενους σε ένα αγώνα για άμεσες και μεγάλες ε, περικοπές. Ε, πολύ κακές εργασιακές συνθήκες που πια αποτελούν τον κανόνα και υποκαθιστούν τις ποιοτικές θέσεις εργασίας. Για την ΤΙΣΑ. Κατά την άποψή μας, οι διαπραγματεύσεις στην ΤΙΣΑ για εμπορικές συμφωνίες αποτελούν μια απειλή για περαιτέρω φιλευθεροποίηση σε αυτόν τον τομέα και περιορίζει τη δυνατότητα του δημοσίου να ρυθμίζει τον τομέα αυτό. Οι ρήτρε όπως η στάνστιλ ρήτρα κάνει πρέπει να μάλλον να αποκλεί περαιτέρω φιλευθεροποίηση και θα πρέπει να εξαιρεθεί αυτό ο τομέας. Θα πρέπει να κάνουμε τα εξής. Όταν έχουμε συζητήσει για, παγκοσμια, για καθολική κάλυψη, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη δυνατότητα ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών όπω αυτέ τι ταχυδρομικές υπηρεσίε. Η Uni Europa και η Uni Globe ε, Europe και άλλε οργανώσει δεν θα ήθελαν να δουν να επαναλαμβάνεται η εμπειρία τη απελευθέρωση του ταχυδρομικού τομέα και να εξάγεται αλλού, γιατί έχει αποτύχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό λοιπόν τα βήματα που θα γίνουν για το μέλλον του ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών καθολικού ε, ενδιαφέροντος, όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με ανοιχτό και διαφανή τρόπο σε δημόσια φόρα ώστε να επιτρέψει στους καταναλωτές, στις οργανώσεις και στους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζί με τους ε, πολιτικούς απελευθέρωση που είχαμε μέχρι τώρα απέτυχε στο να βοηθήσει την εφαρμογή του δημόσιου συμφέροντος στον τομέα αυτό. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι κλειδί σε αυτό το τομέα, επειδή ο τελευταίος λόγος στην Ήπειρό μας είναι δικό σας. Εσείς τον έχετε. Κατά την άποψή μας, οι διαπραγματευτές της ΤΙΖΑ χρησιμοποιούν αυτό το καθεστώς εμπορίου ώστε να δεσμεύσουν τις χώρες σε άγραφη ελευθεροποίηση που διασφαλίζει τις, ε, τα κέρδη των επιχειρήσεων εις βάρος των εργαζομένων και των καταναλωτών. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ακούσει, να εισακούσει αυτές τις ανησυχίες. Δεν θα πρέπει να αποτελεί αυτό σκοπό η οι υπηρεσίες αποτελούν ένα κύριο σημείο, σημείο κλειδί των οικονομιών μας και η φιλελευθερωποίηση, η εμπορική, υποσκάπτει τους τομείς αυτούς, υποσκάπτει τα συμφέροντα των εργαζομένων και των καταναλωτών. Θα ήθελα να καταλήξω λέγοντας ότι δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι η απελευθέρωση των υπηρεσιών δεν αποτελεί μια απειλή. Νομίζω ότι το σώμα σας έχει συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες που είχαμε μέχρι τώρα με την οδηγία για τους εργαζόμενους στο ταχυδρομικό τομέα, οπότε σας ζητάω τώρα το εξής, να μου πείτε το εξής. Αν είχαμε στην ενιαία αγορά ε, δυσκολίες για να εφαρμόσουμε εργασιακή και κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά τους εργαζόμενους σε αυτό το τομέα, πώς περιμένετε να εφαρμόσουμε διεθνεί κανονισμούς μέσω εμπορικής συμφωνίας τη στιγμή που ξέρουμε ότι ήδη αντιμετωπίζουμε σοβαρές δυσκολίε εδώ στην Ήπειρό μας. Και προχωρώντας παραπέρα και κλείνω, θα ήθελα να πω ότι βεβαίως είμαστε υπέρ μιας πλήρους και διεξοδικής εξαίρεσης των δημοσίων υπηρεσιών Άκουσα προηγουμένω με προσοχή αυτά που είπε ο Μάρκο, δηλαδή την ανάγκη να προσδιορίσουμε και να γνωρίσουμε καλύτερα τι επιχειρήσει, τι δημόσιε και τι υπηρεσίε τη ε, κοινοφελού χαρακτήρα. Θα πρέπει να βρούμε ένα νέο μοντέλο δημόσια χρηματοδότηση αυτή τη υπηρεσία. Εμεί θεωρούμε ότι η διάταξη που αφορά τι δημόσιε υπηρεσίε είναι ένα δικαίωμα που έχουν οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να επαναλάβω ότι η φιλελευθερωποίηση και η ολέθρια επίπτωσή της δεν θα πρέπει να εξαχθεί ως καλό μοντέλο, στατικό μοντέλο στον υπόλοιπο κόσμο τη στιγμή που έχουμε, δει τις καταστροφές που έχει επιφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και θα ήθελα τώρα να καλέσω τον κύριο Σάλμπα από την ΕΚΟ να σχολιάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω Είμαι πεπισμένος ότι είναι ε, βασικό στοιχείο ε, ε, η υπηρεσία στην ΤΙΣΑ Και αυτό καλύπτει διάφορα κεφάλαια, παραδείγματος χάρη το εγκάρισιο για τις νομοθετικές ρυθμίσεις, δεύτερον στα τομεακά κεφάλαια και τρίτον στην πρόσβαση στην αγορά. λόγω των οικονομιών κλίμακας και των διασυνοριακών συναλλαγών διαπιστώνουμε ότι οι υπηρεσίε είναι ένα από τα βασικότερα τμήματα των διαπραγματεύσεων. Για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαπραγματεύσεις διότι υπάρχουν διάφορα προσκόμματα που θα επηρεάσουν και το πόσο φιλόδοξο θα είναι αυτό το κομμάτι της συμφωνίας. Υπάρχουν κάποια βασικά προβλήματα στις διαπραγματεύσεις για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Πρώτον, λόγω της κρίσης έχει διαβρωθεί η θέληση να αντιμετωπίσουμε τους διεθνείς φραγμούς που υπάρχουν σε αυτό τον τομέα. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Τα διάφορα μέρη της ΤΙΣΑ δεν έχουν την ίδια, τον ίδιο βαθμό ανάπτυξης στο Πακιστάν και στο Περού, στη ΣΥΠΑ, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε το ίδιο επίπεδο ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ε, μία νομοθετική ρύθμιση σε μια υποκατηγορία χωρών μπορεί να φανεί ότι υπονομεύει το πρότυπο της πολυμερούς διαπραγμάτευσης κυρίως επειδή ε, η Κίνα, η Ινδία παραδείγματο χάρη δεν συμμετέχουν στην ΤΙΣΑ αλλά μετέχουν στην ομάδα εργασίας του G20 για αυτό το θέμα θέμα επίσης ε, για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ε, η ρύθμιση σχετίζεται με τις εθνικές διατάξεις ε, για την χώρα υποδοχής παραδείγματος χάρη και οι χώρες υποδοχής δεν θέλουν να εκχωρήσουν τις αρμοδιότητες που έχουν για τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Ε, δεν θέλουμε λοιπόν να καταλήξουμε σε ρήτρα standstill σε σχέση με τις δεσμεύσεις που μπορούμε να αναλάβουμε. Είδαμε ε, ότι πολλοί υποστηρικτέ αυτής της πρότασης κατέστησαν κοινή ε, δήλωση για να αποτελματωθεί η κατάσταση και να έχουμε μία πρόοδο σε σχέση με τις ρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα και τον οριζόντιο τομέα νομοθετικής ρύθμισης. για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες λοιπόν προς το παρόν δεν προτείνεται ρήτρα standstill αλλά υπάρχει μια προτίμηση για τις εθνικές ρυθμίσεις. Όμως ε, παρόλα αυτά προσπαθούμε να έχουμε μια ελάχιστη ισότιμη πρόσβαση στην αγορά διότι τα περισσότερα μέρη θα πρέπει να αναλάβουν ε, ε, δεσμεύσεις για τις ε, εξωτερικές αλλοδοπές επενδύσεις ή για βασικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στον διασυνοριακό τρόπο παροχής των υπηρεσιών. Για την αναγνώριση, τα μέρη θα έχουν την δυνατότητα να βασίζονται σε μέτρα που έχει υιοθετήσει ένα άλλο συμβαλόμενο μέρος αλλά και για τους παρόχους ε, υπηρεσιών να εφαρμόσουν τις δικές τους διατάξεις η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αναγνωρίζει την ισοδυναμία των ρυθμιστικών καθεστώτων τρίτων χωρών σε αυτό τον τομέα. Τέλος, με αυτές τις διαπραγματεύσεις προκύπτουν διάφορα ερωτήματα που ενδιαφέρουν την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Πρώτον, πόσο φιλόδοξα είναι η συμφωνία για την πρόσφαση στην αγορά, σε ποιο βαθμό τα ε, σχέδια schedule των άλλων μέρων ε, θα ε, εξακολουθούν να εξυπηρετούν τα θετικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, ρυθμιστική πειθαρχία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Πώς εξασφαλίζεται η ισότιμη ώρα ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν κατά της διακριτικής μεταχείρισης και της επαχθούς διοικητικής διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα προαγάγουν και την μελλοντική νομοθετική ρύθμιση. Στη συνέχεια, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική προστασία των δεδομένων. Ε, είμαι σίγουρος ότι θα ασχοληθεί ιδιαίτερα η κυρία Ρέντινγκ με αυτό το ζήτημα. Τέσσερα, αναγνώριση της, του καθεστώτος τρίτης χωρίς για την Πέμπτον, σχέση της ΤΙΣΑ με την ΤΙΤΙΠ, αυτό είναι κέρια σημασία για την ΕΚΟΝ, εφόσον προς το παρόν η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της TTIP δεν επιθυμεί ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Για ποιο λόγο ε, επιθυμεί να συμπεριληφθούν διατάξεις μέσα στην ΤΙΣΑ. Η απάντηση που θα δώσουμε θα πρέπει να συνδυαστεί με τις υποχρεώσεις διαφάνειας που υπάρχουν στο χρηματοοικονομικό κανονισμό. Αυτά. Ε, όλα τα μέλη ε, FSB ε, όπως η Κίνα και η Ινδία πώς μπορούν να αναλάβουν ικανοποιητικές δεσμεύσεις και πώς ε, στα διεθνή φόρα μπορούμε όπως το G20 τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την ΤΙΣΑ μόνο ε, κατά τομέα και κατά βούληση, ε, στη συνέχεια αποκάλυψη πληροφοριών, δημοσιοποίηση πληροφοριών. Αυτό μας ανησυχεί. Αυτό το κεφάλαιο για τις χρηματοδοτικές υπηρεσίες ε, πότε θα σταθεροποιηθεί και πότε θα αποκαλυφθεί στο κοινό, πότε θα δημοσιευθεί. Αυτά. Ε, που μόλις ανέφερα είναι τα ζητήματα που ε, απασχολούν την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και ελπίζουμε να μας δώσετε ικανοποιητικέ απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε για τα συμπεράσματα της Επιτροπής Έκονα, ο κύριος Κόχ από την Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που με προσκαλέσατε ε, να εκπροσωπήσω εδώ την Επιτροπή Μεταφορών. Μα ικανοποιεί η φιλόδοξη ατζέντα της ΤΙΣΑ για την πρόθεση των επιθετικών συμφερόντων της Ένωσης. Το ίδιο σημαντική είναι η διαφάνεια της θέσης της Ένωσης. Ε, πρωτοφανής και μας ικανοποιεί πολύ. Τομείς σημαντικοί όπως οι μεταφορές, όπως ο τουρισμός. Εκεί οι υπηρεσίες παίζουν τεράστιο ρόλο. Το ίδιο ταχυδρομικές και εφοδιαστικές υπηρεσίες εκτός από τους διάφορους τρόπους μεταφορών συχνά πρόκειται για μια αγορά που υποτιμάται και που έχει ωστόσο μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό ιδίως σε εποχές του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο μπορούν να προσφερθούν εκεί νέες υπηρεσίες αλλά και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά για να κλείσουμε κενά στην υφιστάμενη αγορά σε ό,τι αφορά καινοτομία, ευελιξία, το ίδιο για τα διάφορα τις μεταφορές πακέτων, επιστροφές πακέτων κλπ. Εκεί υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες και διερωτώ αν δεν θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες να κλείσουν τα κενά. Το ίδιο σημαντικό είναι να θέσουμε ερωτήσεις τώρα και για τη γεωγραφική κάλυψη και για τις καθολικές υπηρεσίες ε, και απομακρυσμένων περιοχών που δεν πρέπει να μείνουν εκτός ε, σχεδιασμού. Είναι απαραίτητη τόσο και, ένας και μια οικονομική και κοινωνική συνοχή με την διατήρηση των θέσεων εργασίας και ούτω καθεξής και τους κανόνες που διέπουν την κοινωνική συνοχή. Η συμφωνία ΤΙΣΑ δεν επιτρέπεται να ε, οδηγεί στην κατάρρευση των υψηλών κοινωνικών προδιαγραφών. Εμεί της Επιτροπής Μεταφορών έχουμε αρκετή αυτοπεποίθηση για το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρεσβεύει μια ε, λογική απελευθέρωση. η δέσμευση για την καθολική υπηρεσία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί και στον, και στον ε, χώρο, στο πλαίσιο της ΤΙΣΑ δηλαδή, ως αντίθετη με τον ανταγωνισμό, εφόσον περιορίζεται να καλύπτει τις πραγματικές βασικές ανάγκες των χρηστών της. Γι' αυτό αναμένω μια συγκεκριμενοποίηση του ορισμού της καθολικής υπηρεσίας. Χρειάζεται ωστόσο αγώνας κατά των καταχρήσεων των μονοπωλίων. Αυτό είναι σωστό. Το ίδιο χαίρομαι για την ανεξαρτησία των ε, ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Φιέλνερ. Ε, Αγγλικά. Ευχαριστώ. Λίγο σουρεαλιστική μου φάνηκε η συζήτηση παρακολουθώντας ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είμαστε εδώ εν τέλει ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός σε όλο τον κόσμο και η μεγάλη ανησυχία εδώ είναι, ανησυχούμε δηλαδή για μια επιχείρηση που μπορεί, ε, ότι μιλούμε εδώ για, για μια συμφωνία που μπορεί να ανοίξει τον τομέα των υπηρεσιών. Και εδώ λέμε, α, πρέπει να βγάλουμε εκτός αυτόν τον τομέα, εκείνο τον τομέα και ούτε, θα, θα, φτάνουμε, θα φτάσουμε να γίνουμε σαν ελβετικό τυρί στο τέλος, όλο τρύπες, εάν ε, ερμηνεύω σωστά τα αισθήματα που εκφράζονται εδώ. Α, έχει καλή γεύση λέτε το ελβετικό τυρί. Ναι, αλλά όχι οι τρύπε. Εγώ θέλω να κρατήσουμε το τυρί, όχι τι τρύπε. Γι' αυτό, στο πλαίσιο αυτό, να απαντήσω σε μια ερώτηση που τέθηκε για το MOD 4 και αν αυτός είναι προβληματικός ή όχι. Έχουμε ήδη πρόβλημα με την εφαρμογή της οδηγίας για την απάσπαση των εργαζόμενων σε αυτό το mode 4, ακόμα και αν φτάσουμε στην πιο φιλόδοξη ολοκλήρωση της, σύμβασης, της συμφωνίας, δεν θα είναι καν πλησίον της ελευθερίας διακίνησης εργαζομένων που έχουμε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέχουμε πολύ από αυτό λοιπόν. Και γι' αυτό είναι μάλλον ρητορικού χαρακτήρα παρά πραγματικό ρεαλιστικό πρόβλημα στα πλαίσια της ΤΙΣΑ. Θα ήθελα να πω ότι ένα πράγμα που πρέπει να εξετάσει η παρούσα Επιτροπή και γνωρίζω ότι η κυρία Ρέντινγκ το πράττει αυτό, ε, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δηλαδή, είναι οι μεταφορές δεδομένων. Έχουμε και έχω συνεργαστεί εγώ ε, με την άκτα, για, για την περίπτωση της άκτα δηλαδή, έχουμε ε, και πολλά θέματα. Όταν μιλούμε, αυτό δεν είναι επιθετικό ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πολλές υπηρεσίες διαδικτύου και πρέπει να έχουμε υπόψη όταν μιλούμε για τη μεταφορά δεδομένων, δεδομένων μιλούμε για την οικονομία του διαδικτύου αλλά και η παλαιά οικονομία το ίδιο εξαρτάται από μεταφορές δεδομένων διεξήγαγα μια συζήτηση ε, με τον ε, αυτοκινητοβιομηχανία Volvo από τη μικρή μου Σουηδία Μάλλον μου λένε δεν είμαστε πια απλή βιομηχανία, είμαστε βιομηχανία παροχής υπηρεσιών, διότι πάνω το 50% είναι αυτή, αυτή η δουλειά μας. Υπάρχουν πολλές ε, βιομηχανίες που ε, κυρίως τους απασχολούν τώρα οι υπηρεσίες. Μάλλον θα χαρίζανε και τα φορτηγά του αρκεί να ε, υποφελούνται από τον τομέα της προσφοράς υπηρεσιών. Πώς μπορούμε να τους διευκολύνουμε λοιπόν. Γνωρίζω ότι εδώ στην Επιτροπή μας τίθεται κάποια θέματα σχετικά με τον ιδιωτικό χαρακτήρα, αλλά μπορεί να μην έχει τόσο σημασία, αυτό, προστασία των δεδομένων δηλαδή, για τις μηχανές των φορτηγών αυτοκινήτων. είναι δύσκολο να ξεκαθαρίσει κανείς πού πάβει η προστασία των προσωπικών δεδομένων και αρχίζει η προστασία των ε, δεδομένων για τις μηχανές των φορτηγών αυτοκινήτων. Αλλά κάπως πρέπει ε, να δούμε που βρίσκονται τα όρια αυτά και να μην εξετάζουμε μόνο το Google αλλά και άλλα τμήματα της μεταφοράς δεδομένων. Ευχαριστώ εσείς τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Είχα συγκεκριμένη ερώτηση αλλά να πω και το εξή. Για το θέμα των εργαζομένων, αυτό αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία τους μέσω της συνθήκης της Ένωσης. Να το θυμόμαστε λοιπόν αυτό όταν μιλάμε για εμπορικές υπηρεσίες διασυνοριακά. Γιατί κυρίως έχουμε να κάνουμε με τη διεθνή διάσταση των εργαζομένων και της κινητικότητάς τους στην Ένωση. Αυτά που λέμε λοιπόν δυστυχώς δυσχεραίνουν το να υπάρχει διαφανής και ανοιχτή συζήτηση και είναι σημαντικό να υπάρχει τέτοια συζήτηση για την πραγματικότητα και να μην προσπαθούμε να την καλύπτουμε και να την συγκαλύπτουμε. Το ίδιο και άλλους εργαζομένους που έρχονται στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίζουμε την τήρηση των της εργατική νομοθεσίας, της συλλογικής συμβάση και όλες τις άλλες ε, προδιαγραφές. Δεν έχουμε μόνο δηλαδή τα εξωτερικά συμφέροντα της Ένωσης, τα επιθετικά. Είναι σημαντικό λοιπόν να το αναγνωρίσουμε. Αυτό που ήθελα πάντως να ρωτήσω, το οποίο με απασχολούσε από το πρωί, και στις παρουσιάσεις του κυρίου στον και του κυρίου Μπόλους είναι σαφές ότι έχουμε ένα θέμα ως οικονοπίες υπηρεσιών με την πρόσβαση στις αγορές των ΗΠΑ και τα πλαίσια τους. Και αυτό βεβαίως είναι τμήμα των αδιαπραγματεύσεων που έχουμε στα πλαίσια του TTIP. Εμένα το δικό μου το ερώτημα, το εσωτερικό, είναι τι θέλουμε πρώτα. Είναι καλύτερα να επικεντρωθούμε στι διαπραγματεύσει για τι υπηρεσίε στα πλαίσια του TIP και να πετύχουμε εκεί μια σωστή πρόσβαση για τι τηλεπικοινωνίες, τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει κτλ. ώστε να έχουν πρόσβαση στην αγορά ώστε να έχουμε ε, μια ισορροπία στο χρηματοοικονομικό κεφάλαιο στη, στο TIP. ή θα το κάνουμε πιο περίπλοκο προχωρώντας μέσω της και ΤΥΠ ταυτόχρονα. Δεύτερον, για τη χρηματοδότηση και εδώ υπόσχομαι να σταματήσω. Έχουμε πληθώρα εμπορικών συμφωνιών. Και ο κ. Μπόλς όμως είπε κάτι ενδιαφέρον να διασφαλίσουμε δηλαδή στο ότι δεν θα καταλήξουμε με πολλές μικρές ε, συμφωνίες οι οποίες είναι ασύνδετες μεταξύ τους, με κενά. Έχουμε ε, έντονους ε, παράλληλους διαλόγους για τα χρηματοπιστωτικά οπότε αναρωτιέμαι ε, ποιο είναι το σωστό μέρος για να γίνει αυτή η συζήτηση Βασιλεία 2, 3. Θα μείνει εκτός αυτό. Πώς σχετίζονται αυτά μεταξύ τους. Γιατί αρχίζει να περιπλέκεται η εικόνα αν τη δούμε τομεακά και αν δούμε τις ε, εμπορικές συμφωνίες και τη συνεργασία όσον αφορά τα αριθμιστικά ζητήματα διεθνώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, και σου Ναι, ε, μια ερώτηση για την Επιτροπή στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων TTIP όπου στο θέμα των υπηρεσιών υπάρχει σύνδεση με την ΤΙΖΑ. Η Κομισιόν λοιπόν ρωτάει και ζητάει από τις ε, μέλη να επανεξετάσουν το κατάλογο 2 και να επανεξετάσουν τις ε, επιφυλάξεις τους για το θέμα των υπηρεσιών. Η Κομισιόν λοιπόν μας είπε μ, πόσο προσπίζεται την ενιαία έτσι, εικόνα και το νέο δόγμα για τις ευρωπαϊκέ υπηρεσίε. όμως ζητά από τις χώρες μέλη να μειώσουν τις απαιτήσει τους όσον αφορά ε, το θέμα των υπηρεσιών. Ναι, ευχαριστώ. Τώρα οι περιγνώμονές μας. Θέλετε να σχολιάσετε τα σχόλια που ακούσατε. Τρία λεπτά ο καθένα από εσά. Και στο πρώτα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να πω δύο-τρία πράγματα σε λιγότερα από τρία λεπτά. Καταρχάς, για την κινητικότητα των εργαζομένων. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. Εμείς συνεργαζόμαστε με τα συνδικάτα για να διαπραγματευτούμε πολιετής συμφωνίες. Έχουμε επιτυχημένες τριετής συμφωνίες, συλλογικές δηλαδή διαπραγματεύσεις με τους εργαζομένους μας. Βεβαίως, έχουμε και την οδηγία η οποία προχωράει. Αλλά το μεγαλύτερο θέμα που αφορά νομίζω κυρίως εσάς είναι το κοινό στα προσόντα και κοιτούν διάφορες χώρες ε, και οργανώσεις το πώς θα μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν αυτό. Και υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίε ε, στο Νέο για την πρόσβαση τώρα στη ΣΥΠΑ, θαυμάσια αγορά, και η μεταφορά δεδομένων από και προς είναι βεβαίως κρίσιμη αλλά έχουμε μια συμφόρηση ας πούμε πρόσβαση στη τοπική αγορά των ΗΠΑ και το οποίο μας απασχολεί και βεβαίως έχουμε και την παράλληλη συνέχεια των διαπραγματεύσεων στο TTIP. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτά τα δύο ως διαδικασίες αλληλό στηρίζονται ή θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε χωριστά. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπόρος. Ευχαριστώ πολύ για το Mode 4, μια σύντομη παρατήρηση. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τις επιχειρήσεις παροχής οικονομικών υπηρεσιών και τις ανομιλικές συναλλαγές και την οδηγία. Ε, έχουμε το θέμα, ας πούμε, τη συμφωνία με Σιγκαπούρ, Σιγκαπούρ, Λονδίνο, μεταφορές εκεί. Τέθηκαν δύο ζητήματα προηγουμένως από ένα ομιλητή για το TTIP. Από ό,τι βλέπω, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι ασύμβατες οι διαδικασίε TISA και TTIP. Η φιλοδοξία της TISA όσον αφορά ε, το ρυθμιστικό θέμα των χρηματοοικονομικών ε, είναι περιορισμένες. Γιατί είπα, εκτός από τις εθνικές ασφάλειες όπου υπάρχει πρόσβαση και ξέρετε αυτό είναι και μέρος του προβλήματο για το TTIP. Η πρόσβαση στη ΣΥΠΑ και την αγορά τους δεν είναι προβληματική, υπάρχει συνεργασία. Αυτό που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και τα δύο και το ΤΙΖΑ και το ΤΟΤΙΠ είναι οι άλλες χώρες, ας πούμε η Ταϊβάν, ε, τι θα κάνουν αυτές και τις ε, δικές τους ε, ενέργειες, ε, κεφάλαια, καταθέσεις κτλ. Δεν νομίζω να υπάρχουν πολλές μη συνεπείς μεταξύ τους διατάξεις. Το τίτι πάντως είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην ουσία αφορά ακριβώς αυτή την ε, ρήτρα στατστιλ η ΤΙΖΑ αφενός και το ρυθμιστικό κομμάτι του, του Υπάρχουν φραγμοί, αλλά το TTIP είναι σημαντικό για τις οικονομίες μας, ώστε να μειώσουμε τα κόστη. Είναι καλό για το τομέα των χρηματοοικονομικό, για την ε, χημική βιομηχανία κλπ. Ευχαριστώ. Ο κ. Θοδωράκης. Ευχαριστώ. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Σας εύχομαι καλή τύχη στο να, προσ... να, προστατεύσετε τα συμφέροντά μας στις διαπραγματεύσεις στην... στο μέλος από την Επιτροπή των ε, Μεταφορών. Είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε βοήθεια. Πάντως για το Mode 4 ε, δεν θα απαντήσω γιατί αναφέρθηκα συνάδελφοι προηγουμένως το ε, τομέακα. Ε, για μας, για το τομέα των υπηρεσιών μας, αυτό δεν μας ανησυχεί. Αυτό που ανησυχεί το τομέα των τεχνικών υπηρεσιών και τη της είναι το επίπεδο αριθμιστικής συνεργασίας. Δεν είμαι εμπειρογνώμονας, οπότε δεν θα τολμήσω να αναφερθώ στις νομικές διαφορές μεταξύ της και της Δηλαδή, ποια από τις δύο συμφωνίες προέχει, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Θα έλεγα όμω ότι αν αφαιρέσουμε τη δυνατότητα των ΟΤΑ και των εθνικών κυβερνήσεων να ρυθμίσουν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, τότε το συμφέρον των πολιτών και των εργαζόμενων το αφήνουμε στα χέρια των επιχειρήσεων και των διαπραγματευτών. Και αυτό από τη σκοπιά των συνδικάτων ένα παράδειγμα. Ευχαριστώ. Ναι. Και από την σκοπιά ε, των βουλευτών το ίδιο. Έχει όρεξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει κάτι για την TTIP και την ΤΙΣΑ. Ναι, επιτρέψτε μου να πω πως η επιχειρηματολογία του κυρίου Μπόλς ε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα μέλη της ΤΙΣΑ ε, είναι πολλά και διαφορετικά σε σχέση ή μάλλον ε, είναι διαφορετικά σε σχέση με το βαθμό ε, ανοίγματο ε, της πρόσβασης και μιλώ και για χώρες αλλά και για κατηγορίες, ομάδες χωρών. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Και έτσι, ενδεχομένως στη ΔΙΣΑ θα έπρεπε να έχουμε κάποια βασικά πρότυπα ε, που ε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ως τον πω γιατί και εκεί είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση ανάλογα με τις χώρες δύο μέρη με το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης, ε, την ίδια λεπτομέρεια ως προς τις ε, ρυθμίσεις, ε, το ίδιο επίπεδο ανοίγματος της αγοράς μπορούν ενδεχομένως να βελτιώσουν την, την ρυθμιστική του συνεργασία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ευχαριστούμε. Και τώρα η μόνιμη συγκήτρια, η κυρία Ρέντινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι Μιλώ και εξ ονόματός σας όταν ε, ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση. Ήταν ε, πολύ χρήσιμη η συζήτηση, αλλά είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας και όχι το τέλος. Ε, θα πρέπει να επεξεργαστούμε πάρα πολλά ζητήματα. Θα ήθελα ειδικότερα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Επιτροπή ε, Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Μεταφορών. Θα μας βοηθούσε πολύ να μας δίνατε το κείμενο της παρέμβασής σας. Συνοψίζοντας, ε, διαπιστώνω ότι είναι δύσκολο να κάνω μια περίληψη όλων αυτών των σημείων που τροφοδοτούν τη συζήτηση. Θα ήθελα να πω πως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Σεπτέμβρη του 2014 μέχρι σήμερα μας ενημερώνει με πάρα πολύ ικανοποιητικό τρόπο για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή όσοι εκπροσωπούν τις πολιτικές ομάδες λαμβάνουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Ήθελα να το πω αυτό διότι όλοι αναφέρθηκαν στο θέμα της διαφάνειας και της πρόσβασης στα έγγραφα των διαπραγματεύσεων. Χρειαζόμαστε πρόσβαση Επιθυμούμε να έχουμε την πρόσβαση και θέλω να τονίσω πώς όσοι εμπλέκονται ε, στις διαπραγματεύσεις αναρωτιούνται γιατί δεν είναι δημόσια τα έγγραφα διότι δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε δημιουργούνται υποψίες ε, όταν παραμένουν απόρριτα κάποια έγγραφα με δημόσια έγγραφα μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό γιατί δεν θα ευσταθούν πλέον αυτές οι υποψίες που εκφράζονται. Κάτι άλλο που ανέφεραν επίσης οι συνάδελφοι είναι πως υπάρχουν τόσες πολλές συμφωνίες που κανείς δεν ξέρει τι ισχύει τελικά. Με τους εμπειρογνώμονες για τη βοήθεια της Επιτροπής μπορούμε να κάνουμε μία συνολικότερη ανάλυση των συμφωνιών που τώρα διαπραγματευόμαστε, δηλαδή να διαπιστήσουμε αν υπάρχουν ε, αντικρώμενα σημεία ή σημεία σύγκλησης, να γίνει ε, μία ανάλυση τόσο ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή, μία ακολουθία ανάμεσα στις διάφορες διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή. Όλοι οι ομιλητές επίσης αναφέρθηκαν στο ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια καλή συμφωνία η οποία μπορεί να είναι πιο περιορισμένη από ό,τι ελπίζουμε, αλλά θα είναι αποτελεσματική, διότι οι εμπορικοί φραγμοί εμποδίζουν την δραστηριότητα των επιχειρήσεών μας και ταυτόχρονα οι αξίες, οι αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διαφυλάτονται. Αυτή είναι μια σύνοψη της συζήτησης. Το πιο σημαντικό, Πρόεδρε, είναι να δούμε ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε τώρα. Δηλαδή, η λίστα του ντου. Τι πρέπει να κάνει εφ' εξής η Επιτροπή. Να δει τις συζητήσεις, ε, τις συμφωνίες ε, που τώρα ε, διαπραγματευόμαστε, για την ΤΙΣΑ θα λειτουργήσουμε ε, με τίσιο ρυθμό, δηλαδή θα συνεχίσουμε τη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και τους εμπλεκόμενους φορείς. Θα διοργανώσουμε ακροάσεις για ειδικά ζητήματα. Η ροή των δεδομένων είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό, Πιστεύω να συζητηθεί, το Mode 4 επίσης και κάποια άλλα επιμέρους ζητήματα. Πιστεύω, Πρόεδρε, πως καλό θα ήταν να συνθούμε και με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων για αυτά τα θέματα, να διοργανώσουμε μια κοινή ακρόαση με εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και κατά τη διάρκεια του 2015 να συντάξουμε μια διακομματική έκθεση ούτως ώστε να συμβάλλουμε στις διαπραγματευτικές εντολές από πλευρά του Κοινοβουλίου πρωτού λήξει το 2015 και εφόσον εσείς ασχολείστε πρόεδρε με τον, ε, την TTIP συγκεκριμένα μόλις ολοκληρώσετε μπορούμε να αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε το θέμα τίσα. Προς τους συναδέλφους από την Επιτροπή ΕΚΟΝ και Τρανς ε, θα ε, έλεγα ότι θα συζητήσουμε και πάλι τη συμβολή σας και θα απευθυνθούμε και σε άλλες επιτροπές διότι χρειαζόμαστε και τεχνικές αλλά και πολιτικές ε, συμβουλές. Αυτό θα έχει καθοριστική σημασία. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε κυρία Ρέντινγκ. Νομίζω ότι αναφερθήκατε στα βασικότερα σημεία των μελλοντικών μας εργασιών και εστιάσατε την προσοχή σας και σε κάποια ε, ειδικότερα ζητήματα. το δεύτερο ήμιση του 2015 θα πρέπει να γίνει γνωστή η θέση του Κοινοβουλίου και ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για τη διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στις διάφορες ε, διαπραγματεύσεις. Στη γάμα Δέλτα Trade σίγουρα θα έχετε ένα πίνακα που δείχνει τη διασύνδεση όλων αυτών των διαπραγματεύσεων. Θα μπορούσατε ενδεχομένως να μας δώσετε το υλικό που έχετε για να έχουμε μια σφαιρικότερη άποψη για όλες τις προϊούσες διαπραγματεύσεις. Πολύ ευχαριστούμε και τους εμπειρογνώμονες. Πολύ χρήσιμη ήταν η ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστούμε που ήρθατε και θα τα ξαναπούμε στις 3.